So, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zur Ausschusssitzung. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε θερμά στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ξεκινάμε σχεδόν στην ώρα μας, διότι έχουμε μια αρκετά φορτωμένη ημερήσια διάταξη και πάλι. Ίσως να αλλάξουμε τα σημεία 20 και 21 και να τα εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα. Ο λόγος για αυτό είναι ότι αν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις ψηφοφορίες νωρίς, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε τα σημεία 20 και 21 της μερισσές διάταξης σήμερα. Ανακοινώσει της Προεδρίας. Για άλλη μια φορά έχουμε πλήρες γλωσσικό καθεστώς. Κροατικά, Μαλτέζικα και Εσθονικά δεν προσφέρονται, λέει ο Πρόεδρος δεν παρέχονται σήμερα και θα κάνουμε μια προσπάθεια να ξεκινήσουμε αυτή την συνεδρίαση. Ξεκινάμε προσπαθώντας να εξοικονομήσουμε χαρτί. Έτσι λοιπόν δεν τυπώσαμε διπλά τις τροπολογίες ώστε να μην στέλνουμε τόνους χαρτιού και μετά να το ανακυκλώνουμε κάναμε, καταστήσαμε διαθέσιμα τα έγγραφα της συνεδρίασης μόνο για του, τα μέλη ή επισκέπτες στις συνεδριάσεις της Επιτροπής θα χρειαστεί να τυπώνουν οι ίδιοι τα έγγραφά τους ή να χρησιμοποιούν το σειρματοδίκτυο και να τα κατεβάζουν στους υπολογιστέ τους έτσι ώστε μέχρι το τέλος ε, μέχρι να έχει ολοκληρωθεί αυτό το μέτρο θα έχουμε εξοικονομήσει 50 τις 100 χαρτιού, 80.000 τόνους χαρτιού. Ελπίζω λοιπόν να γίνει η προσαρμογή μια και καλή και αν τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και περνάμε σε μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Δύο λόγια μόνο, κύριος Μπόκρος. Συμφωνώ απολύτως να εξοικονομούμε χαρτί αλλά όταν ζητάω αγγλική μετάφραση, παρακαλώ μην μου δίνετε την ουγγρική. Τουλάχιστον να γίνεται αυτό που ζητάμε. Ε, Συνήθω ε, είναι γνωστό ότι διανέμονται τα έγγραφα στη μητρική γλώσσα του κάθε βουλευτή, αλλά βεβαίω ε, ευχαριστούμε για την επισήμανση και θα μεριμνήσουμε ώστε να ικανοποιηθεί η επιθυμία σα. Και περνάμε στο σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη, όπου έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΜΑ, τον κύριο Γκουίντο Ράζη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις στο παρελθόν. Μας έχουν απασχολήσει γενικά οι υπηρεσίες οι αποκεντρωμένες. Η Επιτροπή μας είναι υπερήφανη και ικανοποιημένη από, τις, ε, από την ύπαρξη των υπηρεσιών. Φυσικά παρακολουθούμε τη δουλειά σας και θέματα που έχουν να κάνουν, ε, που συζητούνται και που έχουν να κάνουν με συγκρούσεις συμφερόντων, <coughs> παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει δεν καθυστερώ άλλο και για να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας πιο αποτελεσματικά, σας δίνω το λόγο για την παρουσία σας, παρακαλώ. Thank you. Ε, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την πρώτη, για πρώτη φορά ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο για να σχολιάσω την υλοποίηση της νομοθεσίας για τη φαρμακοπαγρύπνηση και να σας πω μερικές σκέψεις για αυτό το πρώτο έτος το οποίο επισήμανε την ανάγκη αλλαγής των δυνατοτήτων μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναγνωρίσω τον προσωπικό ρόλο που διαδραματίσατε πολύ από εσάς ώστε να γίνει αυτή η νομοθεσία πραγματικότητα. Ήθελα επίσης να αναγνωρίσω την αφοσίαση και τη δέσμευση των εμπειρογνωμόνων και του προσωπικού του οργανισμού που εργαστηκαν τόσο σκληρά για πάνω από ένα έτος για την επιτυχία επιτυχή εφαρμόγη της ε, νομοθεσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από μόλις τρεις μήνες, στις αρχές του Ιουλίου 2012. Η νέα Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου της φαρμακο... Επαγρύπνησης, γνωστή ως ΠΡΑΚ, η έβδομη επιστημονική μας επιτροπή έχει συνεδρίασει μόλις τρεις φορές ε, αλλά εργάζεται αυτή τη στιγμή σκληρά εσείς οι νομοθέτες έχετε παίξει το ρόλο σας και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας ωστόσο η πολυπλοκότητα και το μέγεθος ε, του έργου που έχουμε μπροστά μας ε, δεν πρέπει να υποτιμάται Γνωρίζουμε ότι κανένα φάρμακο δεν είναι ποτέ χωρίς κίνδυνο και ότι μόνο η πραγματική χρήση ε, φαρμάκων δείχνει ε, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος ε, ωφελών και κινδύνου και τώρα με αυτή την καινοτόμο νομοθεσία όλα αυτά έχουν γίνει δυνατά. Ωστόσο πρέπει να πω έχουμε ελάχιστη εμπειρία όσον αφορά το χειρισμό εκθέσεων και μηνυμάτων από έναν τόσο μεγάλο αριθμό ετερογενών ε, πηγών όπως οι εκθέσεις ασθενών, ε, οι εκθέσεις επαγγελματιών του τομέα της υγείας, ε, οι εκθέσεις των διαφορών εταιριών και των 27 διαφορετικών χωρών που σύντομα θα είναι 28. Οι προσδοκίες λοιπόν είναι αυξημένες Θα πρέπει να προσέξουμε ακραίες υπερβολικές αντιδράσεις ε, σε συγκεκριμένα συμβάντα και θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε και το αντίθετο, να αποφύγουμε να αποφύγουμε την, ε, το να μην αντιδράμε έγκαιρα. Τώρα θα σας ε, παρουσιάσω μερικούς προβληματισμούς. Μετά από την έγκρισή σε αυτή την Επιτροπή τον Ιούλιο πέρυσι, εγώ έγινε εκτελεστικός διευθυντής ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων τον Νοέμβριο του 2011. Σε αυτό το χρόνο συναντηθήκα με το προσωπικό, τα μέλη της Επιτροπής και τους εμπειρογνώμονες και συνολικά ε, απέκτησα μια σωστή ενδελική γνώση του οργανισμού, του περιβάλλοντος το οποίο δραστηριοποιείται και των ενδιαφερομένων του. Στον οργανισμό ανακάλυψα ότι το προσωπικό και, το και η διαχείριση ήταν αρμόδια και ε, αφοσιωμένα, έτοιμα για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτή η δέσμευση είναι η δύναμη που επιτρέπει στον οργανισμό να παρέχει αποτελέσματα, να αλλάζει, να μεταβάλλεται και να προσαρμόζεται ώστε να διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα του συνεχώ μεταβαλλόμενου περιβάλλοντο στο οποίο εργάζεται. Αυτή η πολυπλοκότητα οφείλεται στην δομή 7 αλληλένδετων επιτροπών, καθεμία με διαφορετικού ρόλου που όλες ε, εξετάζουν τον κύκλο ζωής των διαφορών φαρμάκων από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτή. Η πολυπλοκότητα επίσης οφείλεται στις νέες θεραπευτικές ευκαιρίες, νέες τεχνολογίες, ε, νέες συστήματα παροχής ε, φαρμάκων, που, χορήγησης φαρμάκων που ορισμένες φορές μας καλούν να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τα φάρμακα. Το περιβαλλον λοιπόν στο οποίο εργάζεται ο οργανισμός θα συνεχίσει να μεταβάλλεται και ίσως ταχύτερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει συνεχώς ε, να είμαστε σε επαγρύπνηση για αυτή την αδιάκοπη διαδικασία αναδιοργάνωσης που θα συνεχιστεί στο μέλλον. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι αλλαγές ε, θα χρειαστεί να έχουμε εμπιστοσύνη και να δυσφαλίσουμε τη φήμη μας. Ε, η εμπιστοσύνη και η φήμη θα εξαρτηθούν ε, από τη σοβαρότητα του οργανισμού μας και από τη διαφάνεια ε, κατά την κοινοποίηση των αποφάσεων. Η όλη διαδικασία είναι απαραίτητο να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής από αυτή την άποψη. Πιστεύω η υποστήριξη της Επιτροπής υπήρξε πολύτιμη. Μας ενθάρρυνε συνεχώς να βελτιώνουμε τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία και την ομοιομορφία των, και τη συνοχή των επιστημονικών μας γνωμοδοτήσεων. Αυτό συνέβαλε σε τεράστιο βαθμό στην αύξηση του επίπεδου εμπιστοσύνη και φήμης Συμπερασματικά είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίζετε τις προσπάθειες του οργανισμού για να τηρήσει αυτές τις αρχές και να οικοδομήσει ε, την εμπιστοσύνη 500 εκατομμυρίων πολιτών. Τέλος, θα θέλω να αναγνωρίσω το συμβολή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, του καθηγητού Νίστικο ε, και Λέμερ. Είναι σημαντικό να θεωρήσουμε αυτού του δύο καθηγητέ ω σύνδεσμο μεταξύ τη Επιτροπή και του οργανισμού και του ευχαριστώ για το έργο του. Από τότε που άρχισα να εργαζόμαι σε αυτόν τον οργανισμό έλαβα γνώση τη υποστήριξης τη παρούσα Επιτροπή ε, στο έργο μα σε διάφορου τομεί. και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη, την επικοδομητική σας ε, συμβολή Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Και τώρα μπορούμε να ακούσουμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Πρώτα θα παρακαλώ την Ντάκμα Ροκ που είναι και η ε, συνάδελφος ε, που έχει την επαφή με την αίμα. Να μας πει λοιπόν τις δικές σας θέσεις. Πολύ συχνά άλλωστε αναφέρεται όχι μόνο στους συντονιστές αλλά και στην Επιτροπή. Κυρία Μάρτροκ, Πέρεντ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ράζη. Και πίνω ριστικό. Ο συνάδελφος που κάθεται εκεί στην άκρη. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του καθηγητού που έπρεπε να έρθει σήμερα διότι η κόρη του παντρεύεται αύριο και δεν ε, ήταν εύκολο να ταξιδέψει μέχρι τις Βρυξέλλες. Εγώ του είπα ότι η προτεραιότητα έχουν πάντα τα παιδιά και τα οικογενειακά θέματα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε τον κύριο Ράση, την πρώτη φορά που τον είδαμε εδώ ε, είχε έρθει να μα παρουσιαστεί ω υποψήφιος εκτελεστικό διευθυντής. Ύστερα από 11 μήνες λοιπόν η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του και να μας πει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εμένα με ικανοποιούν αρκετά θέματα. Καταρχά ότι για άλλη μια φορά υπογραμμίζει ο κύριο Ράζη ότι δεν είναι άμυρα κινδύνου τα φαρμακευτικά προϊόντα. Δεν υπάρχει φαρμακευτικό προϊόν άμυρο κινδύνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη όταν συζητούμε θέματα και νομοθεσία για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Πάντοτε Είμαστε πάνω σε ένα, κινούμεθα πάνω σε ένα πολύ λεπτό στρώμα πάγου και πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με υψηλή φάρμακο επαγρύπνηση. Επίσης, με ικανοποιούν τα όσα είπατε εδώ. Έχω δύο-δυόμιση θα έλεγα ερωτήσεις που φαντάζομαι θα ενδιαφέρουν και τους συναδέλφους ή κάποιους από αυτούς. Αναφερθήκατε στο περίπλοκο έργο της ΕΜΑ, τις επτά αλληλοσυνδεόμενες επιτροπές, επί παραδείγματι. Αυτές οι επιτροπές, η HMP, παραδείγματι, η επιτροπή που ασχολείται με τα φάρμακα για ανθρώπους ή για τα φάρμακα για τα παιδιά και λοιπές επιτροπές τείνουν, όπως βλέπουμε εδώ και στις δικές μας τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, να μετατρέπονται σε μικρές ηγεμονίες και ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση κύριε Ράζη. Αυτές είναι λοιπόν μικρές ηγεμονίες τείνουν να διονγκώνονται και να αναπτύσσουν ένα δικό τους κύκλο ζωής, πράγμα το οποίο δεν με ευχαριστεί πάντα. Αναφέρεστε λοιπόν στην οργάνωσή σας, πράγμα το οποίο βεβαίως και θέλουμε να ακούσουμε και εγώ και οι άλλοι συναδελφοί. Αλλά θα σας παρακαλώ να αναφερθείτε και σε κάτι άλλο που είχατε θίξει στην πρώτη σας επίσκεψη εδώ με την υποψηφιότητα. Είχατε πει ότι νέες, διαδικα... πρωτοβουλίες ή διαδικασίες βελτίωσης θα πρέπει να προβληθούν. Επί παραδείγματι, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες ιδέες. Τι εννοείτε, αυτούς τους 11 μήνες. Ξέρουμε βεβαίως ότι το να, αλλάζει, το να αλλάξει κάτι σε αυτές τις ε, διαδικασίε τι παγιωμένε επί χρόνια, είναι σαν να προσπαθεί κανεί να μεταστρέψει ένα δεξαμενόπλιο. Αλλά είναι μια βραδία δηλαδή διαδικασία. Αλλά μπορείτε να μα πείτε τι έχετε αλλάξει και τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε για την ενίσχυση τη αποτελεσματικότητα, για την ενίσχυση των δικτύων και ιδιαίτερω αυτό που εμένα ενδιαφέρει για να συντονίσετε τις δομές της αίμα, τις δομές που βρίσκονται μέσα στην αίμα καλύτερα για να συντονιστεί δηλαδή η δουλειά των διαφορών επιτροπών καλύτερα. Και ταυτόχρονα θα παρακαλέσω να μου κάνετε κάποιο σχόλιο για τις συγκρούσεις συμφερόντων που ξέρω ότι ενδιαφέρουν πολλούς συναδέλφους εδώ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε συχνά με πολλές αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Χρειάζεται διαφάνεια και θα θέλαμε για άλλη μια φορά να καταστήσετε σαφές τι μπορείτε να πράξετε ώστε να καταλαγιάσετε τις επικρίσεις. Ή τι άλλο για την αίμα. Και επίσης κύριε Πρόεδρε, κύριε Γράζη, χρειάζονται εμπιστοσύνη οι οργανώσεις, αλλά και υπομονή χρειάζονται. Και ξέρω ότι δεν είναι όλοι πάντοτε υπομονετικοί. Αυτό είναι μια ε, αυτοκριτική, γιατί και εγώ δεν μπορώ να πω ότι σεμνήνομαι πάνω απ' όλα για την υπομονή μου. Δεν είναι η πρώτη μου η πρώτη μου, το πρώτο μου προτέρημα, το κύριο μου προτέρημα, ούτε το δικό μου είναι κάποιον άλλον βεβαίω. Αλλά, εν πάση εγώ προσπαθώ, προσπαθώ πολύ να το καταπολεμήσω και να βελτιωθώ. Όπω ελπίζω θα πράξουν και άλλοι. Θέλουμε λοιπόν καλή συνεργασία, στενή συνεργασία με την Επιτροπή μα. Εμεί θα σα υποστηρίζουμε πάντοτε όταν κάνετε καλή δουλειά, διότι ε, μπορεί να μην ήταν πάντοτε ανέφελε οι σχέσει μα, αλλά όλοι νομίζω επιδιώκουμε την τελειότητα. Η πιο στενή συνεργασία μεταξύ τη ΕΜΑ και τη Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τη δικής μας Επιτροπής, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Έχω και άλλους ομιλητές. Θα σας διαβάσω τα ονόματα και μετά κλείνω τον κατάλογο. Γιατί όσοι θα έρθουν από εδώ και μπρο, του άλλου δεν έχουν ακούσει και την παρέμβαση. Äh, Miroslav äh, Nikolasic, dann die Kollegin äh, Kukovic, äh, Bobros, dann Michel Rivasi, Corinne Lepage und dann möchte ich auch noch den Vertreter des Management Boards, dem και μετά θα ήθελα να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Λύση όμως πρώτος. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Ράση για την ε, παρουσίαση εδώ και την ευκαιρία που μας δίνετε για την ανταλλαγή απόψεων. Ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο εδώ, τον παλιό μας συνάδελφο και την Ντάγμαρ. Σύντομα. Διαφάνεια στις κλινικές επαληθεύσεις. Πριν από κάποιους μήνες πήγαμε στο Λονδίνο μια μικρή αντιπροσωπεία και συζητήσαμε την αίμα, σημειώσαμε με ικανοποίηση ότι ε, είναι πολύ δραστήρια η αίμα με στην αναζήτηση της ε, διαφάνειας. Έχει λάβει υπόψη τα αιτήματα τα δικά μας, τα προωθεί, προσπαθεί να βελτιώσει τη διαφάνεια, αλλά βεβαίως πρόβλημα παραμένουν οι κλινικές δοκιμές σε τρίτες χώρες όπου υπάρχει κα... Ε, κακή, χειρότερη προστασία του ασθενούς. Άρα λοιπόν θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες προστασίας για τον ασθενή εν γέννη στην Ευρώπη, αλλά πάνω απ' όλα για τον ε, ε, άνθρωπο εκείνο ο οποίος συμμετέχει ως πείραματόζω σε ένα πείραμα. Στο Λονδίνο λοιπόν το πρόβλημα το οποίο ακούσαμε, μας περιγράφηκε, ήταν ότι τα περισσότερα αιτήματα τα καταθέτουν οι, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και όχι εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν τα θεμητά επιχειρηματικά ή επαγγελματικά συμφέροντα. Ερωτήσαμε λοιπόν πώς μπορούμε να περιμένουμε καλύτερη συμμετοχή και του δημόσιου ε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος περισσότερο στις ε, προσπάθειες αυτές. Αυτό το οποίο με κατέπληξε στην επίσκεψη του Λονδίνου ήταν η λειτουργία των advanced therapy, των προηγμένων ε, θεραπείων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται προϊόντα που δεν έχουν εγκριθεί από το 2007 και μετά και, κάθε, και αυτά είναι η πρωτοπορία βέβαια και η καινοτομία, κάθε μέρα επιχειρήσεις αποστέλουν επιστολές για να πούνε ότι α, η νομοθεσία που ισχύει μας δυσκολεύει τη δουλειά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην καινοτομία, στις ε, νέες εφευρέσεις και ρωτώ τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση για τις επιχείρησεις. Ευχαριστώ κύριε Μακκέβαν. Um, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς κύριε Ράζη που ήρθατε να μας επισκεφτείτε σήμερα. Εγώ θέλω να σχολιάσω κάτι που είπε η Ντάγμαρ σε σχέση με την, Ευρωπαϊ... με την Επιτροπή γιατί ξέρετε όταν ασχολήθηκα με την αναθεώρηση της φαρμακοεπαγρύπνησης της σχετικής νομοθεσίας με εντυπωσίασε το ότι υπήρχαν αδύνατα σημεία πολλά στην νομοθεσία και ήρθαμε σε επαφή με την ε, ΕΜΑ η οποία δεν είχαν εμπλακεί όταν έκανε τις προτάσεις της η Επιτροπή. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες Επιτροπή και αίμα, αλλά εμεί θεωρούμε θα έπρεπε για αυτό το θέμα τα κοινού ενδιαφέροντο να συνεργάζονται. Δηλαδή, τελικά άλλος νομοθετεί, άλλος εφαρμόζει τον νόμο και δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Επομένω θα έπρεπε να σας έχουν συμβουλευτεί. Για την φαρμακοπαγρύπνηση, τη σχετική νομοθεσία, έγινε σημειώθηκε πρώτος, καλό αυτό. Ε, στο Λονδίνο κάνετε εκείνη την ε, συνάντηση. Και ξέρω ότι θα πρέπει για την φαρμακοπαγρύπνηση να δουλέψουμε πιο εντατικά. Και είναι και το θέμα της ενημέρωσης των ασθενών, γιατί αν θυμάστε υπήρχε εμπλοκή στο Συμβούλιο και είχαμε πει να υπάρχει ε, πόρτα στο, στο ίντερνετ και είπαμε ότι αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο, αλλά τέλος πάντων όντως έχετε συμβάλει πάρα πολύ και εσείς και οι εθνικοί φορείς και από αυτού το για πέστε μας είπατε ότι σας προβληματίζει αυτή η ενίχνευση σήματος από την αλλά η αλήθεια είναι αυτό φιλτράρεται από τους εθνικούς φορείς, δεν είναι διαθέτηση στο Λονδίνο και και, και, μαθαίνετε για διάφορους ε, ασθενείς, για διάφορα θέματα ε, φαρμάκων. Ε, αυτό περνάει από τις εθνικές αρχές πρώτα. Άρα... Δεν ξέρω τι κάνετε για να παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα των, των επιμέρους φορέων. Εσείς μπορείτε να κρίνετε πόσο αποδίδουν, τι δουλειά κάνουν, πόσο αποτελεσματικοί και είναι αυτοί οι εθνικοί φορείς. Τέλος δε για την φαρμακοπαγρύπνηση έχω να σας πω ότι υπάρχουν εδώ κάποια θέματα που τα παρακολουθούμε εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για οπωσδήποτε την συζήτηση για τη λίστα των φαρμάκων τη χρησιμοποίηση κάποιων συμβόλων ξέρω ότι έχουν αρχίσει συζητήσει για τα σχετικά σύμβολα και κάποιοι τώρα κάνουν λόμπι κατά αυτού του μέτρου. Μετά όμω από όλα αυτά τα σκάνδαλα με τα φάρμακα, μετά από όλα έχουμε δει, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτό ακριβώς αφορά η αναθεώρηση που θέλουμε να γίνει, που ξεκίνησε πέρσι. Και άρα θέλουμε του, του χρόνου ήδη να έχει ξεκινήσει αυτό το σήμα και να υπάρχει το σύμβολο αυτό πάντως σε όλα τα φάρμακα. Ευχαριστώ κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε και Διευθυντή, ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που αναφέρατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις ότι θα παραμείνετε σε στενή συνεργασία με την παρούσα Επιτροπή που είναι η κύρια Επιτροπή όσον αφορά θέματα υγείας και φάρμακα και ιατροτεχνολογικές συσκευές. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι πρακτικό. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια νέα κατάσταση, νέα εμπιστοσύνη, νέες επιτροπές, νέα άτομα στην αίμα και εξαιρετικό είναι όλο αυτό και όπως είπε ο θα χρειαστεί και κάποιος χρόνος για να γίνουν όλα αυτά. Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρετε με τρόπο επωφελή για τους ε, ασθενείς και με εξαιρετικά τελικά αποτελέσματα. Αυτή είναι φυσικά η γνωστή αρχή την οποία εγώ υποστηρίζω πλήρως. Το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Σε ορισμένες ε, περιπτώσεις, όπως έχω ακούσει και όπως με έχουν ενημερώσει από διάφορες χώρες, ορισμένοι εμπειρογνώμονες που είχαν ας πούμε επαφές με φαρμακευτικές εταιρείες ως ε, εμπειρογνώμονες, γιατροί, ε, ερευνητές μπορεί να εξετάστηκαν από 7 επιτροπέ τη ΣΕΜΑ ή μπορεί να βρίσκονται σε επιτροπέ ΣΕΜΑ ενώ είχαν ίσω επαφέ με ε, ε, φαρμακευτικές εταιρείε παλιότερα ενώ νέοι διπλωματούχοι είναι αρκετά καθαροί εντό εισαγωγικών ώστε να μην υπάρχει θέμα διορισμού του στι επιτροπές σα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πολύ απλή. Πώ αποφασίζετε ποιο είναι επιλέξιμο και ποιο δεν είναι. Υπάρχει δυνατότητα να ορίστε κάποιον που δεν θα είναι μέλος των επιτροπών σας αλλά συνεργάτης εάν έχει ήδη κάποια εμπειρία στον κόσμο της φαρμακευτικής και με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ευχαριστώ. Κουκοβιτς. Κύριε Κουκοβιτς. <clears throat> in uh, lepo pozdravljen in dobrodošel. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Ράση εδώ. Και να επισημάνω ότι τα φάρμακα πάντοτε ενέχουν κινδύνους. Και έτσι εδώ τίθεται το πρώτο μου ερώτημα. Τον έχω έναν ασθενή που πάσχει από χρόνια νόσο Πώς μπορώ να συνδυάσω διαφάνεια και πάγια επικοινωνία με τον ασθενή αυτό ταυτόχρονα. Ώστε όταν προκύψει ένα νέο φάρμακο, να είμαι βεβαίως, βέβαια, ότι μπορώ να το αξιοποιήσω και να βεβαιωθώ ότι είναι κατάλληλο για τη θεραπεία του, του κάνει καλό. Διαφάνεια δηλαδή στην εισαγωγή δύο ισοδυνάμων φαρμάκων. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να εξασφαλιστεί και θα ήθελα βεβαίως να σας προστηρίξω ότι, στην ιδέα ότι θα πρέπει όλοι οι ειδικοί να ε, συμβάλλουν στην αξιολόγηση των ε, φαρμάκων. Και όταν κυκλοφορεί ε, ένα φάρμακο στην αγορά, τότε θα πρέπει και τα ονόματα αυτών των ειδικών να καθίσετε γνωστά να το έχουν υποστήριξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Μπόγκρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τη σήμερα ημέρα η Ευρώπη θεωρείται μία από τις ε, περιοχές του κόσμου όπου ε, δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες για ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης όμως όσον αφορά τη φραγμοβιομηχανία και τα σχετικά ακόμα ε, είμαστε πρώτο πρωτοπόροι και όντως εκεί υπάρχουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Το ερώτημα το δικό μου είναι Πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα, ούτω ώστε να αποκτήσουμε και άλλα πλεονεκτήματα για να ξεπεράσουμε τα σύνορα της Ευρώπης. Άρα σας ρωτώ πώς ακριβώς συνεργάζεστε με διάφορου φορεί εκτός ε, ευρωπαϊκών σύνορων, τόσο ώστε να προωθήσετε αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Και βέβαια εκτός αυτών πώς μπορούμε να ωφελήσουμε γενικότερα όλο τον κόσμο. Κύριε Μπλάζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ορίζουμε τον κύριο Ράζη σε αυτή την Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που ο κύριος Ράζη έχει αντιληφθεί το γεγονό ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Τον ευχαριστώ για αυτό λοιπόν. Ταυτόχρονα όσον αφορά τα προβλήματα συγκρούση συμφερόντων έχουν, γίνει, έχουν σημειωθεί πρόοδοι. Ωστόσο, αναρωτιέμαι για την παρακολούθηση, για το follow-up. Καλό είναι να έχουμε όλε τι δηλώσει ε, των εμπειρογνωμόνων, αλλά πώ παρακολουθούνται όλα αυτά και ποιε κυρώσει μπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση μη τηρήση των διαδικασιών. Ταυτόχρονα είχαμε την περίπτωση του κ. Λόγκρεν, ο οποίος ε, έφυγε, που είχε κάποιο, ανήκε σε κάποιο ιατρείο. Ναι, ωραία, έχουμε ωραίες προδιαγραφές, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχουν κυρώσεις. Εάν κάποιος φύγει από την αίμα, όπου είχε μια θέση ευθύνη και πάει κάπου όπου έχει συμφέροντα και αυτό σχετίζεται με την αίμα, ποιες είναι οι κυρώσεις για αυτά τα άτομα. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πως θα αποτρέψουμε άτομα που έχουν αναλάβει ευθύνε ε, στην αίμα να πηγαίνουν μετά να βρίσκουν δουλειά στην φαρμακευτική βιομηχανία. Εάν δεν υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις πηγαίνουν τελικά γιατί εκεί κερδίζουν χρήματα. Το δεύτερο όσον αφορά τις κλινικές μελέτες. Είχαμε ζητήσει οι κλινικές μελέτες να βρίσκονται στο διαδίκτυο διότι διαφάνεια σημαίνει δημοσίευση όλων των στοιχείων. Ε, κάτι τελευταίο για τα φάρμακα επανειλημμένως ε, είδαμε προβλήματα όσον αφορά τις παρενέργειες των φαρμάκων. Αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι υπάρχουν επαρκείς μελέτες ώστε να ορίσουμε κάποια φάρμακα ως προβληματικά και να τα βγάλουμε από την αγορά. Όσες φορές υπάρχουν αμφιβολίες ρίχνετε τις ευθύνες στους γιατρούς, προειδοποιώντας ουσιαστικά τους γιατρούς. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο καθαροί θα έπρεπε να γνωρίζουμε σε συνάρτηση με τις μελέτες πώς θα αποσύρουμε ορισμένα φάρμακα, πόσες μελέτες χρειάστηκαν για το Mediator, για το εκείνο το εμβόλιο που προκαλούσε αναρκοληψία, πόσες μελέτες είχαμε. Εμένα το πρόβλημά μου είναι πώς γίνεται η ειδοποίηση και πότε. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω ως πρόταση σε σχέση με τις πρόοδους που έχετε σημειώσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μήπω θα ήταν σκόπιμο να οργανωθεί μια ομάδα εργασία με βουλευτές όπως εδώ ας πούμε από την Επιτροπή από τη δική μας Επιτροπή με όλου τους ευσυνείδητου βουλευτές που έχουμε εδώ που θα μπορούσαν να παρακολουθούν ε, ας πούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου τα προβλήματα με την απαλλαγή θα θέλαμε λοιπόν να δούμε περισσότερου βουλευτέ σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω μετά όσα είπε η συναδελφός μου, κυρία Ριβάζη, και να δηλώσω την ικανοποίησή μου για τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα που λάβατε σε σχέση με τις δυσκολίες που συνάντησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Αυτός ο έλεγχος των δηλώσεων συμφέροντος, η διασταύρωση των διαφόρων συμφερόντων στον οργανισμό και σε εθνικό επίπεδο επέτρεψαν να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να δηλώσω την ικανοποίησή μου και να σας συγχαρώ. Πιστεύω ότι περισσότερο από ποτέ στη δύσκολη κρίση που περνάει η Ένωσή μας σήμερα οι πολίτες χρειάζεται να μας δείξουν εμπιστοσύνη και τα ζητήματα υγείας είναι το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα που μας απασχολεί μετά από τα ζητήματα απασχόλησης. Συνεπώς η εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε όλοι στον οργανισμό σας αποτελεί παράγοντα ε, εξισορρόπησης γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω αφορά το follow-up, την παρακολούθηση, αναρωτιέμαι ουσιαστικά το τι θα συμβεί τώρα. Κάποιο συναδελφό μου ρώτησε ποιου εμπειρογνώμονε θα χρησιμοποιείτε και πώς θα λειτουργείτε. Δηλαδή πώς οι σωστοί κανόνες πρακτικής σας μεταφράζονται σε πραγματικές αποφάσεις που θα λάβετε και σε πραγματικές νομοδοτήσεις που θα παράσχετε. Πρόκειται να κάνετε εμπειρογνωμοσύνη αντιφατική, δηλαδή για κάθε θέμα μάλλον που θα παρουσιάζεται θα υπάρχουν οι θέσεις υποστήριξης και οι αντίθετες θέσεις, η απόψη υπέρ και κατά. Θα συνεργαστείτε και με εμπειρογνώμονες ε, που θα μπορούσαν να δώσουν μια καθολική άποψη του θέματος εντός και εκτός της βιομηχανίας θεωρείτε ότι οι αποφάσεις που θα χρειαστεί να λάβετε μπορεί να αλλάξουν κατεύθυνση έχοντα, μεριμνώντας διαρκώς ε, για την υγεία των πολιτών γιατί παρότι είστε ένας ε, ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγχεται όχι μόνο τη χρήση των φαρμάκων αλλά και την πρόληψη. Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι δεσμοί με τους υπόλοιπους οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εργάζονται στον τομέα της πρόληψης. Οι ασθένειες κοστίζουν πολλά στην Ευρώπη παρότι η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας μας. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε καλύτερες μεθόδους πρόληψης ώστε να μειωθούν οι, παθολογίες, οι ασθένειες ε, και η χρήση φαρμάκων και να παρέχουμε καλύτερη ζωή στους πολίτες. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Περίλο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ παρεμβαίνω σχεδόν τελευταίος ε, πρώτον για να χαιρετήσω τον πρόεδρο Ράση που ε, διορίστηκε πολύ πρόσφατα τον Νοέμβριο του 2011 και πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε το έργο που καλείται να πράξει ένας οργανισμός αυτού του τύπου. Ε, είπατε ότι τα φάρμακα δεν είναι χωρίς κινδύνους. Έτσι λοιπόν τα καθήκοντα που σας ανατίθενται είναι όλο και πιο δύσκολα. Αφετέρου εγώ σκέφτηκα ότι η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών που ουσιαστικά εποφελούνται από τις πρωτοβουλίες της ΕΜΑ η υγεία λοιπόν αυτών των πολιτών εξαρτάται πραγματικά από τις δράσεις αυτού του οργανισμού. Ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και γι' αυτό παρενέβην Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος της Καλαβρίας όταν ο συνάδελφος εδώ ήταν πρόεδρος της περιφέρειας και ήθελα να σας πω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και είμαι βέβαιος ότι η παρουσία του με υψηλό κύρος και το αντιλήφθηκα σήμερα το πρωί γιατί είδα και το είδα και από τη συντονίστρια μου τη Μακέβαν. Είδα λοιπόν ότι παρουσιάζεται αυτή με υψηλό κύρο λόγω της τεράστιας επιστημονική του εμπειρία, ε, στα φάρμακα θα συμβάλλει σημαντικά στις, ε, στις σημαντικές πρόοδους της ΕΜΑ. Θυμάμαι ότι όταν ήταν πρόεδρος περιφερειάρχης τότε θέσπισε τη σχολή, τη φαρμακευτική σχολή στο Καταντζάρο και τότε μου ανέθεσε να κόψω την κορδέλα μαζί με τον ε, πρόεδρο της σχολής ε, ε, Επιτρέψτε μου λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να αναφερθώ, για αυτή την εξαιρετική σχέση που είχα μαζί και εύχομαι ε, τα καλύτερα για το έργο του εκτελεστικού διευθυντή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις προσωπικές παρατηρήσεις που κάνουν πιο ζωντανές στις συζητήσεις μας. Και είναι καλό να ακούγονται τα εγκόμια για τη δουλειά που έκανε και στην Καλαμβρία και βέβαια εδώ ο συνάδελφος Τώρα ας ακούσουμε τον συνάδελφο, κύριο, τον πρώην συνάδελφο, κύριο Νηστικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριο Όλοι τώρα αντιλαμβάνονται γιατί γιατί, γιατί θα είμαι τόσο κολακευμένο ε, για τόσο συναρπαστική θεωρώ την ε, επίσκεψη αυτή. Ευχαριστώ εσά, ευχαριστώ την ώρα του Μπέρντ. Ε, είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα φυτικά, φυσικά φάρμακα. Ήμουν ε, ο δημιουργός και εκείνη δημιουργός, α το πούμε, έχω την πατρότητα, εκείνη τη μητρότητα εκείνη στις έκθεσεις και, ο Πίτερ Λίζε, οπότε βλέπετε τώρα πόσο σου δίκιο είχαμε όταν δώσαμε για τα κύτταρα, για του αγώνες εκείνους. Γιατί το Νόμπελ, είδατε που πήγε φέτος για τον επαναπρογραμματισμό των κοιτάρων αυτών, οπότε βλέπετε με πόση χαρά παρίσταμε εδώ και δεν μπορώ να ευχαριστήσω και τον Μάριο Πυρίλο. Μάριο ήσουν καταπληκτικός αντιπρόεδρος, αλλά επίσης θα πρέπει να σας πω την άποψή μου για τον ρόλο του καθηγητού Ράζι. Ξέρετε, είναι φοβερή οι προκληθούς φοβεροί που μπορεί να τρέμουν τα χέρια κάποιοι που ασχολείται με αυτή τη δουλειά την τόσο δύσκολη, την τόσο περίπλοκη. Και εγώ, ξέρετε, έχω συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβουλίο του ΣΕΜΑ και βλέπετε πρόκειψε μια νέα, ένα νέο στρατηγικό όραμα, περισσότερος δυναμισμό, σε αυτή την δραστηριότητα αυτό το οποίο χρειαζόταν ήταν να υπάρξει συντονισμό μεταξύ των επιμέρους διαφορετικών επιτροπών που ασχολιόντουσαν με αυτή την επιστημονική πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και πάρα πάρα πολύ καλά τα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θα πρέπει να προσθέσω ότι για την φαρμακοεπαγρύπνηση την ώρα το τότε που κάναμε την έκθεση είχα κατεβάσει, γίνει την τροπολογία και είχαμε πει για την αρχή της πρόληψης οπότε κάθε φορά που τίθεται σε εμπορία ένα νέο φάρμακο το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τότε η εταιρεία οφείλει να συμβάλλει στην ε, έρευνα. Στη σήμερα μέρα υπάρχει φαρμακοπαγρύπνηση και ναι, είναι αλήθεια, είναι δύσκολη η καιρή, δύσκολο να, να, βρεθούν πόροι, όμως, όμως μια μικρή επιβάρυνση είναι θεμητή. Θα πρέπει επομένω οι ε, εταιρείε φαρμάκων με κάποιο μικρό ποσό να συμβάλλουν. Το πρόβλημα όμως είναι να βρει κανείς Ντάγμαρ την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης του να λειτουργεί έτσι αυτό το σύστημα και ότι, του ότι δεν χρειάζεται να φτιάξουμε ένα νέο αίμα, ένα νέο οργανισμό φαρμάκων μπορούμε να έχουμε τη φαρμακοπαγρύπνηση, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, μπορούμε να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις σε όλους όσοι ανησυχούν για τα τοξικά, για τα πολλές φορές μοιραία αποτελέσματα χρήσης κάποιων φαρμάκων ή κατάχρησης. Κάτι άλλο που παρακαλώ να με βοηθήσετε και, και όλοι εδώ και εσύ όσον αφορά το, την κλινική πλευρά των πραγμάτων ήδη υπάρχει υπάρχει αυτός ο οργανισμός φορμάτων. Με αυτά ασχολείται τόσα χρόνια. Γιατί να έχουμε επικάλυψη. Γιατί να έχουμε κάποιον που να κάνει την ίδια δουλειά σε επίπεδο επιτροπής. Αναπόφευκτα θα έχουμε συγκρούσεις στο μέλλον. Τα έζησα αυτά. Ο οργανισμός CHMP αποτελεί την επιστημονική αυθεντία. Άρα δεν μπορεί να παρεύει κανείς. Προσοχή επομένως για να μην έχουμε σύγκρουση στο μέλλον. Εν κατακλείδη έχω να σας πω ότι είναι βέβαιος πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων με την εποπτεία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής θα μπορέσει να εξισορροπήσει το τι χρειάζεται να λάβει υπόψη και να εκφράσει αυτά τα οποία χρειάζονται οι ασθενείς. Ο Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για το έργο που επιτελέσατε στο Διοικητικό Συμβούλιο και τώρα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ράζη για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί. Ελπίζω να απαντήσω πλήρως. Προσπάθησα να κρατήσω σημειώσεις, οπότε ζητώ συγγνώμη αν ξεχάσω κάτι. Θα προσπαθήσω, αν ξεχάσω κάτι, να το καλύψουμε στη συνέχεια. Πρώτα το ερώτημα της κυρίας Ροτμέρεντ που αφορά την πολυπλοκότητα και το τι κάνουμε ουσιαστικά για να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα και να βελτιώσουμε την απόδοση μας, τα αποτελέσματά μας Ουσιαστικά ακολουθούμε δύο γραμμές, την επιστημονική και την διοικητική. Η επιστημονική γραμμή αφορά τις δραστηριότητες των εμπειρογνωμόνων και των επιτροπών. Όπως γνωρίζετε έχουμε επτά επιτροπές, όπως προείπα. Αυτές οι επιτροπές ε, εξετάζουν διαφορετικά, διαφορετικές πτυχές των προϊόντων. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ένα επιστημονικό συντονιστικό γραφείο που συγκεντρώνει τους πρόεδρους όλων των επιτροπών ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα να προβλεφθούν τα προβλήματα και να υπάρχει συνοχή στην όλη αξιολόγηση μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Αξιολόγηση γιατί μερικέ φορέ ε, οι διαφορέ διαγραμμάτων, υπάρχει χρονική διαφορά δύο ετών μεταξύ επιτροπών. Προσπαθούμε λοιπόν να παρέχουμε κάποια σταθερότητα και συνοχή στι δραστηριότητε και στι αποφάσει μα. Δεύτερον, ε, έχουμε μια ομάδα επιστημονικών σύντακτων. Αυτή η ομάδα βοηθάει τον εκάστοτε εισηγητή να, να αποκτήσει μια πιο ομοιόμορφη, μια πιο στιβαρή και μια πιο συνεκτική γνωμοδότηση που θα είναι ε, εύκολο να γίνει κατανοητή όταν ε, ληφθεί η απόφασή μα, διότι η κοινοποίηση, η ενημέρωση βασικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ε, Ένα από του σημαντικότερου παράγοντε οικοδομή εμπιστοσύνη. Η τρίτη δράση έχουμε... Είχαμε μέχρι σήμερα 76 ομάδες εργασίας ε, με τη συμμετοχή 3.500 εμπειρογνωμόνων. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα μπορούμε να ενσωματώσουμε όλες τις γνώσεις που μπορούν να παρέχουν αλλά δεν ευθυγραμμίζουμε ούτε, αν δεν ευθυγραμμίσουμε και δεν οργανώσουμε τη διαδικασία θα χάσουμε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης που μπορεί να μας ωφελήσει και εδώ ερχόμαστε στη διοικητική λοιπόν προσέγγιση έχουμε μια δραστηριότητα που την ονομάζουμε OPEX, Operation Excellence ε, επιχειρησιακή αριστεία ουσιαστικά που αναλύει κάθε επιμέρους διαδικασία. Αυτή έχει αποδώσει ήδη σημαντικά αποτελέσματα με την ε, μεταφορά ατόμων σε άλλες θέσεις, ε, με την απελευθέρωση αποδέσμευση ορισμένων πόρων. Κάποιοι πόροι, κάποια άτομα έχουν ε, αλλάξει, έχουν μεταφερθεί σε άλλα σημεία που χρειάζονται και επίσης έχουμε αποδεσμεύσει και κάποιου οικονομικού πόρους για να ολοκληρώσω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλη η διαδικασία ενημέρωση και τεχνολογίας Όλες οι διαδικασίες ουσιαστικά επικοινωνίας και τεχνολογίας που βασίζονται σε πολύ περίπλοκες βάσεις δεδομένων αυτή τη στιγμή αναδιοργανώνεται εκ βάθρων. Φαίνεται να είναι κάτι πολύ απλό και συνηθισμένο, αλλά μας δίνει μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει σε εμά. Ε, έχουμε αποδεσμεύσει εντός τριών μηνών έτσι 3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διαθέσουμε σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα στη φαρμακοεπαγρύπνηση όπου τα τέλη δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί πυλώνες ε, που μας βοηθούν να έχουμε απόδοση. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τις αντιδράσεις της διοίκησης υποστηρίζουν, μας υποστηρίζουν ιδιαίτερα σε αυτή την προσέγγιση. Ελπίζω λοιπόν αυτό να καλύπτει ένα κομμάτι της ερώτησης, ένα μέρος της ερώτησης. Ο κύριος Φελής ε, ανέφερε το ζήτημα της διαφάνειας. Σύμφωνα με τις σημειώσεις που κράτησα, Έχουμε πολλές δραστηριότητες ε, για τη διαφάνεια. Αποτελεί φυσικά προτεραιότητα για μας. Για παράδειγμα, δημοσιεύουμε τα πρακτικά ε, και τις ημερησίες διατάξεις των επιτροπών. Ξεκινάμε την ΚΟ με την ΠΙΔΙΣΙΟ και την ΠΡΑΚ ε, και θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που θα αποκτήσουμε ώστε το συντομότερο δυνατόν να μπορούμε να δημοσιεύουμε όλες τις ημερήσεις διατάξεις και όλα τα πρακτικά όλων των επιτροπών. Οι κλινικές δοκιμές, τα στοιχεία μάλλον των κλινικών δοκιμών θα δημοσιευτούν σύντομα. Αυτό θα απαντήσει σε μια ερώτηση που έχουμε ακούσει συχνά από πολλούς από εσάς στις 22 Νοεμβρίου θα έχουμε μια σημαντική συνάντηση στην οποία θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να παρέχουμε ουσιαστικά τα στοιχεία και πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι ουσιαστικά μόνο οι ανταγωνιστές μας που θα λαμβάνουν αυτά τα δεδομένα αλλά να τα δημοσιεύουμε με τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να καταλαβαίνει πώς αυτά τα στοιχεία τεκμηριώνουν τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Ελπίζουμε να βρούμε μια ισορροπία βάσει το συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων σε αυτή την άσκηση δημοσίευσης των κλινικών στοιχείων, την οποία ελπίζουμε να υλοποιήσουμε στα τέλη του έτους. Όπως είπατε, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ισορροπίας μεταξύ των αυτών που εποφελούνται και αυτών που εκμεταλλεύονται με αρνητικό τρόπο τα δεδομένα. Τώρα όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, έχουμε υλοποιήσει πολλές δράσεις. Τον Απρίλιο του 2012 ε, κυκλοφορήσαμε ένα έγγραφο προβληματισμού για την αποδοχή αποτελεσμάτων δοκιμών ή δοκιμών που έρχονται εκτός Ευρώπης. ουσιαστικά για να εξασφαλίζεται η υλοποίηση της δήλωσης του Ελσίνκη, της διακήρυξης του Ελσίνκη. Και φυσικά οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις θα αποτελούν μεγάλο κομμάτι αυτής της άσκησης. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα περιορισμού των εξουσιών των επιθεωρητών μας. Ε, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε απευθείας για ηθικούς λόγους πώς οι ασθενείς εκτός Ευρώπης ε, ουσιαστικά συμμετέχουν στις δοκιμές και καλούνται να συμμετέχουν στις δοκιμές. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Ελπίζω πραγματικά να μου δοθεί ευκαιρία να το εξετάσω όλο αυτό με προσοχή και να δούμε και τις νομοθετικές πτυχές. Τι δηλαδή ε, βοήθεια, υποστήριξη μπορούμε να προσφέρουμε γενικότερα. Τώρα όσον αφορά τις προηγουμένες θεραπείες, Οι προηγούμενε θεραπείε αποτελούν σημείο ανησυχία για μένα, διότι στην προηγούμενη δουλειά μου πραγματοποιούσα έρευνε σε προηγούμενε θεραπείε. Συνεπώ, ελπίζω, έχω ελπίδε για αυτέ. Σήμερα σημειώνεται μια επιτυχία, η πρώτη γονιδιακή θεραπεία στον κόσμο. Πολύ ίσως πιστεύουν ότι δεν ήταν επιτυχία λόγω του πόσο δύσκολη ήταν η λήψη μιας τελικής απόφασης ε, αυτή η γονιδιακή θεραπεία ε, για δύο χρόνια ουσιαστικά συζητήθηκε σε, ε, συζητήθηκε σε δύο επιτροπές και εν τέλει βρέθηκε μια λύση με συγκεκριμένες υποδείξεις θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που έγινε αξιολόγηση με μια πλήρω εντελώς διαφορετική προσέγγιση εκτός από το στατιστικό εργαλείο που είναι το πρωταρχικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε εκτός από τον αριθμό ε, δράσεων πρέπει να δούμε λοιπόν τη θετική πτυχή το γεγονός ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας νομοθεσίας δέσμευση των επιτροπών να συζητούν επάπειρον μέχρι να βρουν τη λύση και βρήκαν τη λύση ώστε να παρέχουν αυτές τις θεραπείες στην αγορά και να ανοίξουν το δρόμο, ένα νέο δρόμο. Πιστεύω ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό. Μα οδηγεί να γίνουμε πιο θαραλέοι και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις προηγουμένες θεραπείες. Ένα άλλο ε, πράγμα που με κάνει αισιόδοξη είναι ότι αν κοιτάξουμε τι γίνεται με τις προηγουμένες ε, θεραπείες, το 80% των προϊόντων και υπάρχουν νομίζω 250 προϊόντα, είναι αρκετά στις δοκιμές φάσης 1 face 1 to trial όπως λέει ο, ο μιλητής που σημαίνει πολύ προηγμένη φάση μπορούμε να προβλέψουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα ολοκληρωθεί, μέσα στο επόμενο θα ε, ολοκληρωθεί η φάση αυτή και θα έχουμε δοκιμάσει 250 προϊόντα σε ένα πιο έμπιστο περιβάλλον όπου θα έχουμε την ικανότητα να κρίνουμε ε, αυτή την εντελώς νέα προσέγγιση και αυτές τις νέες θεραπείες. Αυτό με καθιστά αισιοδόξο. Επίσης όσον αφορά και την εναλλαγή το μέλλον του προσωπικού στον οργανισμό μου προβλέπω κάποια αλλαγή στην ε, πρόσληψη ε, προσωπικού χρειαζόμαστε τώρα χημικούς ε, ειδικού στη στατιστική που θα μπορούν να αξιολογήσουν τις αποφάσεις και τα στατιστικά στοιχεία. Αυτή είναι στο σύνολο προσέγγισή μας. Σας τα είπα ίσως λίγο συγκεχημένα, αλλά είναι πολλές δραστηριότητες ε, και συνεχίζονται. Κυρία Μακέβεν, Ρωτήσατε για την Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι, ε, για την Επιτροπή, ε, νομίζω ότι η συνεργασία μας ξεκίνησε πολύ όμορφα, πολύ συστηματικά, τακτικά ανταλλάσσουμε απόψεις με τον Γενικό Διευθυντή. Γνωρίζω ότι οι συνεργάτες μου διαρκώς για κάποιες αιτίε ε, βρίσκονται σε επαφή με ε, την Επιτροπή. Ίσως να έχουν... δυσκολευόμαστε λίγο να παρακολουθούμε όλες τις ε, δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον ε, θα αναγνωριστεί η εμπειρογνωμοσύνη μας και θα αποτελέσει κομμάτι της νομοθετικής διαδικασίας τεχνική μας συμβολή ουσιαστικά, τα τεχνικά στοιχεία που μπορούμε να παρέχουμε και οι εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε του καθημερινού κόσμου, του πραγματικού κόσμου, πιστεύω ότι έχουν υψηλή αξία και πιστεύω ότι η Επιτροπή θα τα εκτιμήσει ιδιαίτερα. Αυτή την αίσθηση έχω. Συνεπώς δεν προβλέπω τεράστια προβλήματα για το άμεσο μέλλον. Για αυτό το μαύρο σύμβολο είναι αλήθεια. Η διαβούλευση κράτησε αρκετό χρόνο. Συζητήθηκε, συζητήθηκε και δυστυχώ δεν πρόσωπε το ίδιο των πολιτών. Οπότε θα κάναμε κάποιο εξωτερική διαβούλευση με την ομάδα εργασία και νομίζω ότι τελικά συμφωνήθηκε. Το σύμβολο εγκρίθηκε. Οπότε αυτή τη το θέμα στα χέρια τη Κομισιόν για την τελική απόφαση. Από ό,τι γνωρίζω, αυτή τη στιγμή διεκπεριώνεται. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Θίξατε ένα από τα θέματα που με απασχολούν περισσότερο. είναι θέμα της ε, διαφορετικότητας του, του ετερογενούς ας πούμε μεταξύ ασθενούς ιατρικού προσωπικού που ήταν το, το, πρόβλημα του ιατρικού προσωπικού που είχε να κάνει με την βάση δεδομένων ήταν το ζήτημα του εθνικού συστήματος το πρόβλημα. Είχαμε δηλαδή 27 διαφορετικά ιατρικά συστήματα, τελείως διαφορετικά, οπότε το θέμα ήταν πώς θα γινόταν η ανείχνευση και η περιγραφή του σήματος. Και δυστυχώς δεν υπήρχε η γνώση του πώς θα εκαθαριστεί ούτως υπήν το σύστημα, γιατί ένα από τα προβλήματα θα ήταν ο, ο προαπλασιασμός του σήματος. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε για το ίδιο συμβάν μέχρι και τρία μηνύματα, σήματα. Και αυτό λόγω ακριβώς της ε, ποικιλία που υπήρχε. Και δυστυχώ δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία. προπαρασκευή έγινε, αλλά δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία. Ήδη στο website μας έχουμε τουλάχιστον 100 ενεργές ουσίες που για αυτές έχει ανατεθεί η ανείχνευση και παρακολούθηση στα κράτη-μέλη. Επομένως υπάρχουν ήδη ε, τέτοιες διαδικασίες ανταλλαγής εμπειριών, συνεργασίας, είτε ακριβώ όλοι ενδιαφέρονται για το θέμα. Experts. Οι εξπέρι, εμπειρογνώμονες τώρα. Η διαδικασία επίλυση των συμφερόντων σημαίνει ότι θα έπρεπε να διευρύνουμε ε, τους να μειώσουμε, να μειώσουμε τους 4.000 σε περίπου 3.500 εμπειρογνώμονες και αυτό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και ε, είναι καλό σημάδι το ότι υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα για να επισημανθούν οι συγκρούσεις συμφέροντα. Επίσης υπάρχει και το θέμα, το ότι ίσως ε, τα τρία ή ε, πέντε χρόνια της ε, ασυνέχειας συνεργασία εμπειρογνώμων εταιρεία ίσως είναι πάρα πολύ, ίσως να σταματούσε κανείς να είναι ο ειδικό και επαείων και εμπειρογνώμονας. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους επίσης είναι σημαντικός. Απευθυνθήκαμε και στις εταιρείε είναι πιο πιστική όσον αφορά τους εμπειρογνώμενες είναι και θέμα της αμοιβή, όσο, όσο προχωράει ο καιρός έχουν περισσότερη δουλειά. Άρα να μην καταλήξουμε να έχουμε μη εμπειρογνώμονες να κρίνουν τα προϊόντα. Επίσης για τις ε, ακραία σπάνιες ασθένειες έχουμε μόνο έναν τέτοιο ειδικό. Και τώρα να επανέλθω στο πώς μπορούμε να έχουμε πιο οργανωμένη προσέγγιση. Η κάθε επιτροπή χρησιμοποιεί άλλους ειδικού. Οπότε, για κάθε θεραπευτικό τομέα. Είπαμε να δούμε ποιοι είναι οι ειδικοί και όλες οι επιτροπές να χρησιμοποιούν τους ίδιους. Οπότε να έχουμε μια ομάδα ειδικών και τα πράγματα να είναι ευκολότερα. Επίσης, για να δούμε τις FDA τι κάνουν και ε, πώς δουν και αυτοί να επιλύσουν το πρόβλημα του ανταγωνισμού των ειδικών. Επίσης, πώς θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την Sunshine Act. Δεν είναι δική μας ομαδιότητα, αλλά η φαρμακοβιομηχανία πώς θα δούμε να δούμε τι θα πει. Κυρία Ριβαζή, νομίζω, και κυρία Λαπάζου, μας είπαν σχετικά. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να ελέγξουμε την ε, δήλωση σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε ένα κατάλογο ανθρώπων που μας βοηθήσουν, τους ευχαριστούμε, αλλά δεν έχουμε τους πόρους ούτω ώστε να κάνουμε συνεχή παρακολούθηση. Πάντως αυτή η Σάτσο είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ βοηθάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. ζήτησαν από τι εταιρείε να τους ε, δώσουν τον κατάλογο των ειδικών που ασχολούνται με κάθε δοκιμή και ακριβώς τι συμφέροντα εμπλέκονται. Τώρα, λοιπόν, τώρα έχουμε βάλει πάνω σε μία σειρά. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι που τελειώνει μία και έξω. Και έχει εκφύγει το χειρόνο μας πια η δυνατότητα του να βρούμε την τεκμηρίωση τα έγγραφα με τα οποία θα επαληθευθούν τα όσα πρέπει να ελέγχουν για τη σύγκρουση συμφερόντων. Αξιολογούνται κατηγοριοποιούνται και δημοσιεύονται στο website οι σχετικέ δηλώσει. Οπότε έτσι όποιο θέλει μπορεί να μα βοηθήσει και εμεί να κάνουμε τα σχετικά. Και γίνεται η ενημέρωση τη σχετική ιστοσελίδα. Κύριε Κούκοβιτ, αν κατάλαβα καλά τι είπατε, τι να μπορούμε να κάνουμε για να ενημερώσουμε τους ε, ασθενείς σε σχέση με τα φάρμακα για τις ε, χρόνιες ασθένειες. Να δούμε επίσης ποια είναι η λεπίδραση δύο φαρμάκων όταν χωρίζονται ταυτόχρονος. Πραγματικά είναι κρίσιμο αυτό το θέμα και σε επιστημονικό επίπεδο. Είναι δεδομένες, περιορισμένες οι δυνατότητες να μπορέσουμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι ισχύει κάθε φορά. Άρα, στην πράξη προκύπτει αυτό το οποίο λέμε. Αφού δηλαδή χρησιμοποιεί κάποιος το φάρμακο. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να προλάβουμε τις εξελίξεις. Ε, με αυτό, αυτό με απασχολεί και εμένα. Πώς γίνεται με υπεύθυνο τρόπο να ξέρουμε τον προτέρων και πώς γνωρίζει τον προτέρων ο ασθενή επομένως. Για τα γεριατρικά τώρα έχουμε τη σχετική ομάδα. Λειτουργεί στην υπηρεσία μας. Βέβαια και εκεί δυσκολευόμαστε να του πλαισιώσουμε κατάλληλους πόρους, αλλά αυτό χρειάζεται για το πρόβλημα. για τα γυριατρικά. Έχουμε ταυτόχρονη χρήση φαρμάκων και σιγά σιγά αποκτούμε τη γνώση των αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων. Και έτσι το πρόβλημα προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Τώρα, όσον αφορά κάποιο... Τα, τα, τα εργαλεία, νανοτεχνολογία, γενετική και πώς μπορούμε να έχουμε πολλαπλούς τρόπους ανείχνευσης πρώιμων ενδείξεων και να μπορούμε να έχουμε και ικανότητα πρόβλεψη όσον αφορά την ελληπίδραση των φαρμάκων. Ό,τι πληροφορία υπάρχει την λαμβάνουμε υπόψη. Υπήρχε άλλη μια ερώτηση. Ο κύριος Μπόκρος νομίζω, αν προφέρετε το όνομά σας. Ρωτήσατε για αυτό το οποίο σώθουμε να πετύχουμε σε διεθνές επίπεδο. Πρώτα πρώτα. Προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη επιθεώρηση. Καλύτερο έλεγχο. Όταν έκανα αυτή τη δουλειά στην Ιταλία, είχα συγκροτήσει μια ομάδα ελέγχου, τους είχα στείλει στην Ασία ε, όταν έβγαιναν οι δικοί μας έμπαινε η EMA και όταν έφυγαν οι της EMA του Οργανισμού Φαρμάκων, δηλαδή του Ευρωπαϊκού, μπήκαν οι Αμερικανοί. Αλλά όμως ήταν χιλιάδες αυτά τα οποία έπρεπε να, τα που έπρεπε να ελέγξουμε. Οπότε δεν μπορούμε να πάμε σε όλα και άρα αυτό είναι διασπάθηση των πόρων μας. Επομένως, αυτό το οποίο έχει προτεραιότητα είναι η πραγματική προτεραιότητα και σε αυτό μας υποστηρίζει η Επιτροπή για το να έχουν περισσότερες δυνατότητες σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε διάφορα υπομνήματα, έχουμε διάφορες ε, πιστευτικές συμφωνίες. Υπάρχουν, υπάρχουν όλα τα μέσα και τα χρησιμοποιούμε όλα. Σε συνδυασμό με αυτά που έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε άλλωστε και το ξέσπασμα αυτή τη επιδημία μηνυγίδα τη ΕΠΑ. Οπότε δύο μέρε πριν την του τύπου το τα ξέραμε και μας διαβίωσαν ότι είναι εντοπισμένο για το πρόβλημα. Ήταν θέμα της ε, Αμερικανικής Φερνοκοβιομηχανίας όμως. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκαιρα κάποια πληροφορία και κανεί να προλάβει το συμπίνει το πρόβλημα. Κύριε Ριβαζή, νομίζω ότι μπορέσαμε να απαντήσουμε. Δεν ξέρω, συμπάθατε με κάτι και κάποιον ξέχασα. Κάτι άλλο, το οποίο μας είπατε και θεωρώ ότι με ενδιαφέρει, είναι η ερώτηση το πότε θα ενημερώσουμε για τα κλινικά πειράματα προς όφελος του κοινού και συμφωνώ 100% μαζί σας. Στις 22 Νοεμβρίου θα τα πούμε. Και ελπίζω ότι θα εξυπηρετήσει. Και ότι θα υπάρχουν όλα τα σχετικά δεδομένα. και η κυρία Λαπάζ νομίζω το, το ίδιο είχε ρωτήσει. Επίσης, ρωτήσατε τι γίνεται αν θα υπάρξει δημοσιότητα σε απόσυρση φορμάτων. Νομίζω με την τελευταία τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας αυτό προβλέπεται. Είναι νομοθετική ρύθμιση. Και σε όλα τα κράτη-μέλη προβλέπεται να δημοσιεύεται η, η κάθε αποσύς φαρμάκου η αιτιολόγησή της και να αναλύεται σχετικώς. Πρέπει να ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο και τον ε, κύριο για τα καλά τους λόγια. Ελπίζω ότι δεν θα σα διαψεύσω και απογοητεύσω. Συγχωρέστε με αν κάποιον κάτι ξέχασα. Ό,τι θέλετε, επιπλέον μπορώ να σας το διαβιβάσω. Κύριε Ράζη, δεν νομίζω να ξεχάσατε τίποτα. Ήσασταν πολύ διεξοδικός στις απαντήσεις σας. Μας εντυπωσίασαν. Θα σας ξαναδούμε βέβαια τον αύριο. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει μια άγια πρόσκληση από την αίμα για τους συναδέλφους. Και τους εισηγητές το υπογραμμίζουμε του Κοινοβουλίου οι θύρες της αίμα είναι πάντα ανοιχτές όποτε χρειάζεται μία συμβουλή. Και έτσι. Σας ευχαριστώ. Και δεν ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε πάντα τους καλύτερους ειδικού εμπειρογνώμονες στις ε, υπηρεσίες. Έστω και αν καμιά φορά κινούμεθα επί ξηρού ακμής. Και το καλύτερο επιστημονικά αναζητούμε όπως τώρα και το πιο οικονομικό ως λύση, διαφάνεια που είναι πολύ σημαντική, αλλά και η υλοποίησή της στην πράξη. Γιατί μετά τη διαφάνεια που μπορεί να έχουμε σε ένα επίπεδο ακολουθεί η αδιαφάνεια. Πρέπει λοιπόν και στην υλοποίηση των προτάσεων να ε, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια για τη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και εσά και του συνεργάτε σας για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους από το Management Board, από το ε, Εκτελεστικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και θα παραμένουμε μέσα σε επαφή, Κυρίω βέβαια η κυρία Ροτμπέρεντ. So. Jetzt Και τώρα περνάμε στο σημείο 4 της ημερικής διάταξης. Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ροδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινες κατανάλωσης. Με εισηγήτρια την συνάδελφο Μισελ Ριβαζή, την καλό στα όπλα. Μπορείς να λάβεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω λοιπόν εδώ να σας παρουσιάσω μία έκθεση για πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που ορίζει ε, την προστασία του πληθυσμού ε, ως προς την παρουσία δυναργών στοιχείων ουσιών στο είδωρ για ανθρώπινη κατανάλωση. Μια πρόταση που μας αφορά όλους γιατί ε, θα θίξει θέματα συγκέντρωσης ραδιενεργών ουσιών στο πόσιμο είδωρ, στο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση καλύτερα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε λοιπόν σε ποια νομοθεσία παραπέμπει. Εάν κοιτάξουμε την πρόταση της Επιτροπής, ξέρετε ότι υπάρχει μια οδηγία του 98 η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ρηπογόνων όλων δηλαδή των χημικών ουσιών. Όλος παραδόξω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποσπάσει αυτές τις ραδιενεργέ ουσίες και να τις υπαγάγει στο πλαίσιο Ευρατόμ. Αυτό προφανώς μας αφορά όλους και πρέπει να επαγρυπνούμε. Δηλαδή, ουσίες για λόγου χημικ... Ε, χημικές που μπορεί να έχουν επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία πάνε σε μία νομοθεσία, αλλά τα ραδιενεργά βγαίνουν έξω από τη Euratom ε, έξω και πάνε στη Γιουρότομ, εκεί δηλαδή που εμείς οι ευρωβουλευτές δεν έχουμε κανένα λόγο. Γι' αυτό και σας καλώ λοιπόν να αντιδράσουμε ως προς την επιλογή αυτή την νομοθετική. Εγώ επιμένω αυτές οι ραδιενεργές ουσίες να παραμείνουν στην οδηγία για τα ύδατα του 98 και η αδίποτε προδιαγραφή σχετική με τις ραδιενεργές ουσίες να ενσωματωθεί στην οδηγία για τα έδατα του 98. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε υπαγωγή και να πάμε στην Ευρωτών. Έγινε μια γενική συζήτηση χθε συντονισμού και όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούσαν για την παραμονή στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας για τα έδατα. Αυτά είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη, και θα το δείτε στην πρόταση, αποχωρίζεται η φυσιολογική, η φυσική εκπομπή ραδιενέργειας, γιατί ξέρετε ότι μπορεί σε ορισμένε περιοχές να υπάρχει ράδιο 126, όπως το είδωρο Μπαντουά στη Γαλλία. Φυσική εκπομπή επομένως ραδιενέργειας, για την οποία προβλέπει σχετική νομοθεσία ότι δεν μπορεί να ξεπερνά τόσα μπεκερέλα ένα λίτρο ε, ε, ραδιενεργών φυσικών ουσιών, γιατί ξέρετε ότι είναι φυσικό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ανώδυνο, μη επικίνδυνο. Υπάρχει ραδιενέργεια στη φύση, η οποία όμως είναι επικίνδυνη. Άρα θέλουμε να συγκεράσουμε και τα δύο. Διερωτώ με όμως, μήπως πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, γιατί υπάρχει φυσική ραδιενέργεια, εκπομπή ραδιενέργειας και πρέπει να, μετρείτε, να μετράτε έτσι ώστε να ξέρουμε αν μπορούμε να την μειώσουμε, να, την περιορίσουμε, δηλαδή την παρουσία της στα ύδατα, αλλά υπάρχει και η τεχνητή ραδιενέργεια, η οποία είναι άλλη ιστορία και θα πρέπει να την ε, έχουμε υπόψη γιατί αφορά τα λίματα τάρα την εργαλήματα των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μπορεί να φτάσουν μέχρι ε, βιομηχανικέ εγκαταστάσει. Έτσι λοιπόν, εάν συνενωθούν και τα δύο και υποθεί ότι και οι δύο, τα δύο είδη ραδιενέργεια μαζί σωρευτικά δεν ξεπερνούν τα 2,1 ε, μπεκερέλα, ένα λίτρο κτλ. τότε λένε δεν θα υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Όχι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι αν δούμε σωρευτικά και τα δύο, σιωπηρά υπονοείται ότι είναι αποδεκτή η παρουσία ραδιενεργών ουσιών στο νερό. Ακόμα και αν είναι τεχνητό. τεχνητή παρουσία. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να τα ξεχωρίσουμε. Θα υπάρχει η φυσική 1,2 μισιβέρτ ε, και η τεχνητή που θα είναι πιο αυστηρές οι προδιαγραφές με πιο χαμηλό ε, επίπεδο. Γιατί αν βρούμε ιόδιο 131, κέσιο 137, κοβάλτιο μέσα στο νερό, αυτό υπονοεί ότι υπάρχει βιομηχανική εγκατάσταση που απορρίπτει ραδιενεργέ ουσίε στα ύδατα και πρέπει να γίνει έρευνα. Εγώ πρέπει να σα πω ότι ήμουν υπεύθυνη σε ένα ε, εργαστήριο ραδιοπροστασία. Στι ε, έρευνε λοιπόν στα νερά είχαμε δει κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια, και, αλλά πάνω, ανάντι δηλαδή από το εργοστάσιο, είδαμε ότι τα νερά ήταν ραδιενεργά, ήταν μολυσμένα. Και διαπιστώσαμε από την έρευνα ότι δεν προέρχονταν, όπω είπα, από το πυρηνικό αυτό εργοστάσιο, αλλά από νοσοκομεία που βρίσκονταν στα Νάντι και που ρίχνανε τα ραδιενεργά του απόβλητα, τα ιατρικά απόβλητα, μέσα στα νερά του ποταμού Γαρούνα τη Γαλλία. Και Αυτό που θέλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω είναι οι προδιαγραφέ. Τι προδιαγραφέ για ποιον τι θεσπίσουμε. Οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν τι κοιτάξετε, είναι γραμμένε με ε, ενήλικο υποκείμενο. Το νερό όμω, το νερό δεν αγγίζει μόνο ενήλικε. Και παιδί ενό έτου και παιδί έξι ετών και ενήλικο αφορά αυτή η νομοθεσία. Έτσι λοιπόν η αντίληψη για τη ραδιοπροστασία είναι πάντα να μεριμνούμε για την πιο ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, την κρίσιμη όπως λέμε ομάδα πληθυσμού. Γι' αυτό και έχω κάνει εγώ δικές μου προτάσεις οι οποίες απευθύνονται στην κρίσιμη ομάδα πληθυσμού και θα δείτε ότι αφορά συγκεκριμένα τα παιδιά 12 μηνών ενό έτου. Άρα λοιπόν, εάν οι προδιαγραφέ μου είναι καλέ για παιδιά 12 ετών, δηλαδή η μητέρα μπορεί να δώσει το νερό στον πιμπερόν, το νερό από τη βρύση των πιμπερών για το παιδί του ενό έτου, αφορτιόρι, είναι καλό το νερό αυτό, και κατάλληλο και για τους πιο ηλικιωμένους μέχρι και τους, ε, τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Και εδώ ακριβώς έχουμε τη διαφοροποίηση σχέση με την συνθήκη Ευρωτομ του 1996, γιατί αυτή λέει ότι πάντα σε κάθε πρόταση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, τα διάφορα, οι διάφορες ομάδες ηλικίας. Εδώ η Επιτροπή θα ε, αντιδράσει και θα πει άμα ετσάγονται προδιαγραφές για ενήλικες, πώς προστατεύονται τα παιδιά, τα μικρά, με την ίδια προδιαγραφή. Τρίτη παρατήρηση, αρχή του οριπένων πληρώνει. Στην πρότασή μου. Εάν εντοπιστεί τεχνητή ραδιενέργεια, ο ρηπαίνων θα κληθεί να καταβάλει το κόστος των μέτρων αποκατάστασης, της διερεύνησης και αποκατάστασης της ραδιενέργειας. Δεν θα την υποστεί ο φορολογούμενος. Αυτή είναι η βασική αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Και, τρίτο, και τέταρτο θέμα, ενίσχυση των ελέγχων. Λέγεται Φερρυπίν ότι εάν δεν εντοπίζεται πυρηνική ε, ε, πηγή ραδιενέργεια στην περιοχή στην οποία εντοπίζεται αυτό το πόσιμο νερό κτλ. Δεν υπάρχει λόγο να γίνονται έρευνε για ανείχνευση ραδιενέργεια. Όχι. Η δική μου εμπειρία το αντίθετο υποδεικνύει. Ότι δηλαδή όταν γίνονται, όταν λαμβάνονται μέτρα ε, μετρήσεις μάλλον για το παιδί, για το νερό και χημικές μετρήσεις θα γίνουν και ραδιενέργειας μετρήσεις θα γίνουν και έτσι θα έχουμε ένα επίπεδο ε, αναφοράς και θα εντοπίσουμε ενδεχομένως ραδιενέργεια που μπορεί να προέρχεται και από χωματερή και από ε, πυρηνικό εργοστάσιο και από νοσοκομείο. Και όταν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε την προέλευση, τότε μπορούμε να εισαγάγουμε τα μέτρα. Δεν μπορούμε με μία κουβέντα να λέμε ότι εφόσον δεν εντοπίσετε στην περιοχή πηγή ραδιενέργειας τότε δεν γίνεται μέτρηση ραδιενέργεια. Όχι πρέπει πάντα να γίνεται με τις ενέργειες και άπαξ και ε, ε, βεβαιωθούμε ότι τα έχουμε όλα καλύψει, τότε μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Είναι πολύ σημαντικό, σας υπογραμμίζω, το να γίνει αυτή η αλλαγή. Ε, η δε πρόταση της ε, Επιτροπής για την υπαγωγή στην Eurostat, στην Euratom είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί αν μπορέσουμε να το κρατήσουμε στο πλαίσιο της συνθήκης Λισαβόνας, θα μπορέσουμε να έχουμε εμεί τον έλεγχο. Εάν πάει στην Euratom, εμείς θα έχουμε χάσει πλέον κάθε εξουσία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, γνωμοδοτήσουμε, να παρέμβουμε στην νομοθεσία αυτή. Αυτή είναι η ευθύνη μα ως βουλευτών και στην προκείμενη περίπτωση είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη μας. Ευχαριστώ πολύ για την εισήγηση και τώρα παρακαλώ τους σκιώδης εισηγητές να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Νικολάζης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, thank ονομάζομαι, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα και να πω ότι έγινε μια πολύ καλή συνάντηση προπαρασκευής με την κυρία Ριβαζή, την εισηγήτρια. Σε πολλά σημεία συμφωνούμε, έστω και αν δεν έχουμε 100% ταύτιση απόψεων. Πάντως, στις περισσότερες αρχές, τις σχετικές με το κείμενο αυτό, έχουμε νομίζω σαφέστατη ε, σύμπνευση. σύμπλευση. Η ομάδα μου λοιπόν υποστηρίζει τις προτάσεις κυρίας Ριβαζή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει νομική βάση, ότι πρέπει να αλλάξει νομική βάση, διότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το πόσιμο νερό, το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, είναι το νερό το οποίο πίνουμε εμείς που θα πίνουν τα παιδιά μας και είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα της συναπόφασης και αναφερόμαστε ως νομική βάση στο άρθρο 191 που διαφυλάσσει τη δυνατότητα στην αποφασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές ε, λεπτομέρειες που θα πρέπει να συζητήσουμε, κάποιες, ε, κάποια καινούργια στοιχεία που θα θέλαμε εμείς να εισαγάγουμε, παραδείγματι για το ράδιο. και για το νερό, σε, το εμφιαλωμένο νερό. Κάποιες λεπτομέρειες που θα θέλαμε να εισαγάγουμε με τις ε, τροπολογίες που θα καταθέσουμε. το ζήτημα των προδιαγραφών για ενηλίκους ή για παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί ενδέχεται το νερό της βρύσης, το νερό του δικτύου που χρησιμοποιούμε φεριπίν για να φτιάξουμε το βρεφικό γάλα ή το φαγητό των μικρών παιδιών ενδέχεται να είναι μολυσμένο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα ασφαλείς ότι δεν θα παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία των παιδιών ε, με ράδιο, με κέσιο, ε, με οποιαδήποτε άλλη ε, ραδιενεργό ουσία. Εδώ πρέπει να έχουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Πρέπει να έχουμε ένα λογικό επίπεδο, εφόσον εντοπίζετε τέτοιες ουσίες, ένα χαμηλό λογικό επίπεδο ε, παρουσίαση. Αυτά λοιπόν ήταν επικοδομητικό ο διάλογος, θα συνεχίσουμε για να λύσουμε τα εκκρεμή ακόμα ζητήματα. Με την κυρία Ριβαζή συμφωνήσαμε να κάνουμε μία συνάντηση και με εμπειρογνώμονε. βέβαια όχι έναν μόνο εμπειρογνώμονα, αυτό το υπογραμμίζω, θα έχουμε περισσότερους ε, ειδικού. θα προσκαλέσουμε Φερρυπίν και ιατρό, ο οποίος θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην ε, στον εντοπισμό ζητημάτων ε, σχετικών με το πώς μπορούν αυτές οι ουσίες, με ποιο τρόπο επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου και ιδιαίτερα του παιδιού οι ουσίες αυτές οι ραδιενέργειε. Ή λοιπές ουσίες Αυτά λοιπόν, ένα, ένα χρονικό πλαίσιο για το ε, υλικό αυτό. με την έννοια ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για την έκθεση. Και βέβαια η αρχή ορυπαίνων πληρώνει για μένα είναι πολύ σημαντική, την υποστηρίζω και πρέπει να υποστηρίξουμε, να ενισχύσουμε τους ελέγχους, πρόκειται για όρο εκτερών κάνευ. Ε, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ και τώρα τα Νέσκου εκ μέρους Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τανανσέσκου. Πρώτα πρώτα να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Ριβαζή. Το έργο της είναι αξιόλογο. Πολύ. Πάρα πολύ καλά δομημένο και μας τονίζει το πόσο χρειάζεται να έχουμε αυστηρότερους ελέγχους των ραδιενεργών σε σχέση με το νερό που καταναλώνουν οι άνθρωποι. Και συμφωνώ με την συγκήτρια ότι για να έχουμε ασφάλεια δικαίου, για να είμαστε συνεπείς στο κοινοτικό δίκαιο, όσον αφορά το βιοτοπίδο τους, θα πρέπει όλα να εντάσσονται στο πλαίσιο της συνθήκης. Όλες οι ρυθμίσεις. Επίσης, πάρα πολύ θετική αυτή η διάκριση όσον αφορά το σχέδιο κειμένου για ε, ε, το διαχωρισμό μεταξύ φυσικών πηγών ενέργεια και εκείνων που για του οποίου ευθύνεται ο άνθρωπο και οπότε θα πρέπει να γίνεται πέρα κάποια μνήμα όσον αφορά το πόσιμο νερό. Κάτι άλλο τώρα. Θα υποβάλω σχετικά τροπολογίε για το ότι θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια και όλο ένα περισσότερο διαφάνεια για του καταναλωτέ. Θα πρέπει να έχουν τη σωστή ενημέρωση για τι βαθενεργέ ουσίε και για το πώ έχει η κατάσταση, τι γίνεται για το πόσιμο υδρό στην Ευρώπη. Κατόπιν των εξελίξεων στην ε, Ιαπωνία για το πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα θα πρέπει όποτε έχουμε κάποιο ατύχημα να γίνεται άμεση ενημέρωση. Και να έχουμε και αυτό το τηλεφωνικό κέντρο για την καταγγελία, για την γνωστοποίηση εκτάκτων συμβάντων Έχουμε βέβαια διαφορές στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις μετρήσεις, τις μεθόδους ε, για ε, την Αθηνέρη και το νερό. Οπότε αυτό που σας προτείνω είναι τα κράτη-μέλη να έχουν ένα, ε, ένα ευαγγέλιο, ένα, έναν οδηγό των, των αρίστων πρακτικών. Κάτι άλλο που ήθελα να σας προτείνω είναι ότι να δώσουμε στα κράτη-μέλη δύο χρόνια περιθώριο ώστε να συμμορφωθούν με αυτή την οδηγία και όχι ένα έτος όπως προβλέπει η αρχική πρόταση. Και αυτή η διετία θα δώσει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν όσον αφορά την τεχνολογία και έτσι μπορούν να τροποποιήσουν την νομοθεσία τους. Θα ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, εγώ ευχαριστώ. Το κύριο ε, ο κύριος, ο κύριος, ο κύριος που είναι ο σκιώδης Δεν είναι εδώ. Καλά. Ο κύριος Ζήπα. MEP του, ε, ε, e του 2012. MEP of the year. Συγχαρητήρια. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που με ψήφισαν βουλευτή της χρονιάς. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια και συνεργασία πέραν των κομματικών γραμμών. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να πω πόσο ε, ικανοποιημένο είμαι και από την ε, δουλειά στην Επιτροπή μας, από την πολύ καλή συνεργασία και το πνεύμα που έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Ιρβαζή για την έκθεση. Συμφωνώ πλήρως σχεδόν ως προς το περιεχόμενο με την έκθεσή της και ιδιαίτερα ως προ τι επικρίσεις για τη νομική βάση που προτείνεται ε, εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη με 100% τις ε, παρατηρήσεις και της τη κυρία Ριβαζή. Καταρχά, λοιπόν ε, το, η πρόταση ευρωπαϊκή επιτροπή θα είχε σαν συνέπεια να παραγωνίσει το Κοινοβούλιο και δεύτερον με την επιλογή αυτή οι, οι τιμές οι αξίες δηλαδή οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη για την διεξαγωγή των ελέγχων θα είναι τέτοιες που δεν θα αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που θέλουμε. Τώρα, μία ε, σύγκριση για να δούμε σε σχέση με, την, ε, με τις προτάσεις για το πόσιμο νερό αφενός, το οποίο φυσικά είναι πολύ πιο σημαντικό και κρίσιμο από ότι γενικά το νερό το οποίο χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας, πρέπει να έχουμε πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές και εδώ πρέπει να ορίσουμε ουσίες προτεραιότητας για τις οποίες πρέπει να διατηρήσουμε την, ε, τον έλεγχο για να έχουμε στο δυνατόν πιο υψηλό επίπεδο προστασίας για τον πολίτη της Ευρώπης. Η πρόταση λοιπόν της υπαγωγής του νερού αυτού με τη, των διενεργών ουσιών συγκεκριμένα στο πόσμο νερό στην ε, Eurostat προξενεί τεράστιους, ε, προκαλεί τεράστιους κινδύνους γιατί αφήνει καταρχά τα κράτη-μέλη κάθε ε, περιθώριο για το αν θα διεξεγάγουν ελέγχους, υπό ποιους όρους θα διεξεγάγουν τους ελέγχους κτλ. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον να διανοηθούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν θα, εξασφαλ, δεν θα επιτρέψει να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλείας και προστασίας που χρειαζόμαστε. Πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πιο αυστηροί λοιπόν και να επιστρέψουμε στις προδιαγραφές της προηγούμενης, ε, της, της αρχικής οδηγίας για το πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ε, να αποδέχομαι εγώ την υπαγωγή στην Euro, Euratom αυτής της ε, πρότασης. Η κυρία Ριβασίδε πολύ σωστά λέει ότι θα πρέπει η επαλήθευση να γίνεται και όταν δεν προέρχεται, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για αιτία, για προέλευση δηλαδή ραδιενέργειας. Πρέπει βεβαίως να στοχεύσουμε πάντοτε στην προστασία των πιο ασθενών πολιτών της κοινωνίας μας. Και επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πόσιμο νερό, γιατί δεν μιλούμε για νερό απλώς για ε, γενική ανθρώπινη χρήση, μιλάμε για πόσιμο νερό. Αν φανταστείτε ότι αυτό το νερό μπορεί να το πιει η έγκυος γυναίκα, μπορεί να το πιει το βρέφος, τότε προφανώς θέλουμε πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές από ό,τι έχουμε για τους ενηλίκους. Και εδώ ακριβώς εντοπίζω πολλά κενά της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ ακριβώς χρειάζεται περισσότερη μέρημνα και προστασία. και για τις ε, ουσίες που θα χαρακτηρίζονται ουσίες προτεραιότητας, που θα πρέπει δηλαδή να διερευνώνται πιο συχνά και πιο αυστηρά και να μην ε, επιτραπεί να περνάνε από κάποιο παραθυράκι, πορτούλα, χαραμάδα του νόμου για να ξεφεύγουν του ελέγχου, νομίζω ότι εδώ ιδιαίτερα θα πρέπει να επιμείνουμε. Να μην αφήσουμε τα κράτη-μέλη ελεύθερα στην ε, ε, πορεία αυτή. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί, με πολύ αυστηρούς ελέγχους και επίπεδα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λαπάζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Ήθελα να συγχαρώ την κυρία Συγήτρια για αυτή την πολύ ποιοτική έκθεση. Την υποστηρίζω απόλυτα. Πιστεύω ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το θέμα της ποιότητας του πόσιμου νερού και ειδικότερα ε, η παρουσία τρίτων ουσιών όπως ραδιενεργών ουσιών ε, πιστεύω ότι η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρότι δεν είμαι σκοιοδηση θα υποστηρίξω στην ομάδα στην οποία ανήκω την έκθεση αυτή και τις διάφορες προτάσεις που περιλαμβάνει. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Μέρκης που ήρθε πάλι. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και την εισηγήτρια. Είναι πάρα πολύ σωστή αφετηρία να ξεκινήσουμε την δουλειά μας, να έχουμε καλή συνεργασία και να οδηγηθούμε σε έγκριση αυτού του νομοθετήματος και συμφωνώ όσον αφορά τη νομική βάση. Νομίζω ότι είναι θέμα αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αναπαινθεί στην Euratom. το ποσίμο είδωρο, γενικά η πολιτική για τα ύδατα είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, κυρίως τώρα που το εξετάζουμε σε σχέση με την ε, μόλυνση από ενέργεια. Πολύ σωστά τα λέει εδώ στη δεύτερη Κατοχή του κειμένου της Ευρωπαϊκή Επιτροπής όσον αφορά το εμφιαλωμένο είδωρο κλπ. και θα πρέπει να καλυφθεί φυσικά για το ίδιο το οποίο χρησιμοποιείται για τη ε, βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής. Θα πρέπει να προσέξουμε βέβαια όχι μόνο του ενήλικε αλλά και του αδύναμου κρίκου, στην κοινωνία, δηλαδή του ανηλίκους. Θα πρέπει ομένως να υπάρχει ενημέρωση, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα διαδήματα και έτσι να αντιμετωπίζονται όλοι οι ανακύπτοντες κίνδυνοι. Η συγγήτρια και σκιώδης συγγήτες νομίζω ότι ομονοούν και νομίζω ότι θα έχει έσιο πέρας αυτή η ε, νομοθεσία. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Γιάννσενς από την ε, μονάδα για τη ραδιενέργεια. Ο κύριος Γιάννης, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή εκτιμά το σημαντικό έργο που είχε επιτελεστεί για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Εξετάζουμε πώς θα κάνουμε μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση των πολλών ε, τροπολογιών που προτείνονται. Το κυριότερο θέμα, ωστόσο, είναι η νομική βάση, η συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί για τη συνθήκη Ευρατών που αναφέρεται σε πολλέ από τι τροπολογίε, στα εκτιμώντα και στα άρθρα. Τα επιχειρήματα της εισηγήτριας βασίζονται στην έκθεση Ballot που αφορούσε την αναδιατύπωση της νομοθεσίας 54 αλλά δεν λήφθηκε περισσότερο υπόψη από την Επιτροπή, διότι αφορούσε κάτι περισσότερο από την αδιατύπωση. Θα υπενθυμίσω ότι σε αυτή την έκθεση η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου έκανε ουσιαστικά μια σύσταση. Δεν ε, πήρε αυστηρή νομική θέση όσον αφορά τις αρμοδιότητες η Επιτροπή από την άλλη θεωρεί ότι το κεφάλαιο 3 Υγεία και Ασφάλεια της Συνθήκης ευρωατόμ θα πρέπει να αποτελέσει τη νομική βάση για όλα τα ζητήματα που αφορούν ε, βλάβες προς την υγεία λόγω ραδιενεργών ε, υλικών ή ε, ακτινοβολίας. Αυτό οδηγεί την εισηγήτρια την εισηγήτρια να διαγράψει όλες τις ε, αναφορές στην 96-29. Αυτό είναι δυστυχές και αντιτίθεται στο σχέδιο εκθέσης της Επιτροπής ε, Ήτρε ε, της Judith Merkes, διότι ουσιαστικά μειώνει το επίπεδο προστασίας επειδή παραβλέπει την αρχή ότι θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλά τα επίπεδα όσο είναι εύλογα επιτεύξιμο δεν υπάρχει λόγος ρήπασης ε, στα επίπεδα που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα. Επίσης η εκθέση κάνει τη διάκριση μεταξύ φυσικών ραδιονουκλειδίων και τεχνητών. Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για τέτοιου είδους διάκριση. Ούτε στις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας, ούτε στα τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας. Η διάκριση χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει μείωση των δόσεων ραδιονοκλειδίων λόγω της ανάγκης προσδιορισμού και ελέγχου των πηγών ραδιενεργού Ωστόσο αυτό δεν είναι ο σκοπός αυτής της οδηγίας. Στόχος της είναι η ποιότητα του πόσιμου νερού και όχι ο έλεγχος των ραδιενεργών ουσιών από πυρηνικές εγκαταστάσεις σε νοσοκομεία. Αυτό ο έλεγχο γίνεται βάσει των προτύπων του Ευρατόμ αλλά και στο πρωτογενέ δίκαιο στα άρθρα 25 έω 38 τη συνθήκη Ευρατόμ. Αυτέ οι τροπολογίε λοιπόν πρέπει να απορριφθούν. Ορισμένε από τι προτινόμενε τροπολογίε φαίνεται να έχουν γενική εφαρμογή όχι μόνο για τι ραδιενέργειε ουσίε, αλλά και πέραν των απαιτήσεων ε, της οδηγίας του 98, 1998 χωρίς ε, δικαιολόγηση αυτής της διαφοροποίησης των απαιτήσεων μεταξύ ραδιενεργών ουσιών όπως ε, γίνεται στις χημικές ουσίες. Αυτό σημαίνει όσον αφορά την πρόσβαση της πληροφορίε, όσον αφορά την αρχή πάνω πληρώνει, αλλά και τις τεχνικές απαιτήσεις που προτείνονται στην έκθεση. Άλλο ένα σημείο, χωρίς να μπω σε για όλες τις τροπολογίες, είναι το ποιος θα είναι το άτομο αναφοράς για την αξιολόγηση των δόσεων. Η οδηγία βασίζεται σε μια αξιολόγηση για τον ενήλικα άνθρωπο και βασίζεται σε πρότυπα ασφαλείας ε, ε, όπου πρέπει να εξετάζονται όλες οι ομάδες πληθυσμού διότι σε αυτή την οδηγία ουσιαστικά δίνουμε μια ενδεικτική παράμετρο που καταδεικνύει πιθανά προβλήματα στην παροχή πόσιμου νερού. Αληθεύει ότι για κάποια ραδιονουκλεΐδια, ειδικά τα φυσικά, τα βρέφη έχουν μεγαλύτερο κινδυνό από τους ενήλικες. Αλλά η σπουδαιότητα του κινδύνου της έκθεσης σε, μια τέτοια, σε τέτοιο νερό εκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή και είναι σημαντικό μόνο αν ένα άτομο εκτεθεί υπερβολικά στη ζωή του σε τέτοια επίπεδα ρήπανση. Και ο πρόσθετος κίνδυνος για το βρέφος δεν είναι τόσο σημαντικός από αυτή την άποψη. Το άλλο σημείο που αναφέρεται από την κυρία Ριβάζη είναι ανάγκη ενίσχυση των ελέγχων. Μαζί με όλα τα χημικά και παράβλεψη άλλων πηγών πληροφοριών στο πρωτογενές δίκαιο, όπως ξαναείπα, στα άρθρα 35 και 36 τη συνθήκη Ευρατόμ έχουμε πλήρη παρακολούθηση όλων των ραδιενεργών ουσιών σε όλα τα συστατικά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του ποτάμιου νερού, του ε, υπόγειων υδάτων και του πόσιμου νερού. Αυτό μαζί με γεωλογικέ πληροφορίε, ε, μπορεί να παρέχει να αποτελεί σε επαρκή βάση ώστε να επιχειρηματολογήσει κανεί ότι δεν χρειάζονται ε, πρόσθετη έλεγχοι στο σημείο λήψη του νερού αφού αυτέ τι πληροφορίε είναι ήδη διαθέσιμε εάν δεν υπάρχει πηγή δεν υπάρχει δυνατότητα παραβίαση ε, των προτύπων ποιότητα του πόσιμου νερού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε αυτές τις παρατηρήσει. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη Και τώρα α ξανακούσουμε την εισηγητρία για να κλείσουμε. Παρακαλώ κύριε Ριβεζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για, ε, για τα κύρια σημεία αυτής της έκθεσης, τις κύριες κατευθύνσεις αυτής της έκθεσης. Πιστεύω υπάρχει ομοφωνία στο ότι χρειάζεται να τροποποιήσουμε την νομική βάση. Δυστυχώς όμως η Κομισιόν αντιτίθεται πλήρως. Μα επιτρέψτε μου να σας πω, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν λέτε ότι είναι πιο περιοριστικά τα πράγματα σε επίπεδο ευρατόμ. Αν δείτε τις λεπτομέρειες, αυτό δεν συμβαίνει και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Είναι διανόητο σε σχέση με μια οδηγία για το νερό του 98 που αφορά τις χημικές ουσίες και η οποία αναφέρει ότι πρέπει να μειώσουμε όλες τις καρκινογενείς επιπτώσεις και οι ραδιενεργές ουσίες εντάσσονται εκεί και τις βγάζουμε από εκεί για να κάνουμε μια άλλη οδηγία, αυτό δεν έχει συνοχή. Θέλετε να το περιορίσετε στο πλαίσιο της συναπόφασης με το κοινοβούλιο. Όταν λέτε είναι πιο περιοριστική, ταυτόχρονα όλοι οι κανόνες που δίνονται, όλα τα πρότυπα που δίνονται αφορούν ενήλικες και εσείς ίδια αναγνωρίζετε ότι για ορισμένα ραδιοστοιχεία ο κρίσιμος πληθυσμός είναι τα βρέφη του ενό έτου. Φανταστείτε ότι μιλάμε για το πόσιμο νερό. Εάν υπάρξει ρήπανση στο πόσιμο νερό θα αφορά ολόκληρη τη ζωή ενός παιδιού. Και αυτό που έχουμε μάθει από το Τσέρνομπιλ για τις χρόνιες μολύνσεις, ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα υπάρχουν επιπτώσεις μακροχρόνιες και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Συνεπώς η ανάλυση σα δεν έχει συνοχή. Το τελευταίο, όσον αφορά του ελέγχους, όταν λέτε ότι έχουμε όλες τις πληροφορίες εκ των προτέρων, είναι απίστευτο που λέτε κάτι τέτοιο. Όταν εγώ βλέπω στο Τρικάστα χρειάστηκε ένα ε, περιστατικό για να αντιληφθούμε το πόσο νερό είχε ρηπανθεί εδώ και 20 χρόνια. Η Κομισιόν το γνώρισε ότι υπήρχε μόνιμη μόλυνση με ουράνιο εδώ και 20 χρόνια. Για 20 χρόνια. Κανείς δεν το γνώριζε. Ξέραμε την άλλη περίπτωση ρήπανση με τρίτιο από μια άλλη βιομηχανία. Κανεί δεν το γνώριζε. Δηλαδή, όταν κάνουμε ελέγχου πόσιμου νερού για κατανάλωση από ανθρώπου, πρέπει να ελέγχουμε το σύνολο των ραδιοστοιχείων ώστε να έχουμε ένα σημείο αναφορά. Ελπίζω λοιπόν ότι μαζί με όλου μου του συναδέλφου θα καταφέρουμε πρώτα απ' όλα ομόφωνα να σα πείσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε νομική βάση και στη συνέχεια πιστεύω ότι όλοι μας θα σας καταφέρουμε να σας πείσουμε ότι αυτό που μας προτείνετε δεν προστατεύει επαρκώς τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Το βλέπετε την έκθεση να την συζητήσουμε στις 20 Νοεμβρίου, μάλλον 20 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών και για να αλλάξει η νομική βάση θα πρέπει να περιμένουμε και τη γνωμοδότηση της νομικής επιτροπής η οποία ενδεικτικά αναφέρεται πως ε, θα επιτρέψει να ψηφίσουμε στις 23 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή μας για να πάει μετά στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Αλλά όπως είπα αυτό είναι ενδεικτικό. 23 Ιανουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και μετά Ολομέλεια το Μάρτιο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και τώρα περνούμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίσουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημοσίων συστημάτων ασφάλισης υγείας με εισηγήτρια την κυρία Παρβάνοβα. Παρακαλώ. Thank you, President. Uh, first of all... κύριε Πρόεδρε, πρώτα πρώτα. Καλώ όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή τη και για αυτέ τι βασικέ διατάξει που αφορά τη διατάσταση στην αγορά την φαρμακευτική με τη σημερινή οικονομική συγκυρία θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αρχές οι οποίε κρίνουν την τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα. Τώρα, πριν δούμε τι βασικέ ε, διατάξει τη εκθέσεώ μου, πρώτα-πρώτα να σα υπενθυμίσω περί τίνο πρόκειται και ε, περί τίνο δεν πρόκειται, γιατί στου διαδρόμου κυκλοφορούν πάρα πολλέ φήμε. Θέλουμε εδώ πέρα τώρα κάποια μέτρα διαφάνεια για τι τιμέ των φαρμάκων και για τα συστήματα ασφάλισης υγείας βέβαια. Δεν θέλουμε εδώ τώρα να καλύψουμε ποιος κρίνει την υπολογική πολιτική. Αυτά είναι εθνικές πολιτικές, κρατικές πολιτικές. Ούτε καλύπτουμε την εναρμόνιση των τιμών των φαρμάκων ή για το κατά πόσο να πρέπει να υπάρχει μια, ένας κατάλογος πανευρωπαϊκός. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό σήμερα για την αγορά. Δεν υπάρχει νέα αγορά φαρμάκων στην Ευρώπη. Ούτε επίσης καλύπτουμε την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια των φαρμάκων. Αυτά καλύπτονται από άλλα νομοθετήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φάρμακο επαγρύπνηση και όσον αφορά την επιστροφή των φαρμακευτικών εισόδων θέλουμε να υπάρχει ε, αποτελεσματικότητα. Άρα θα σας πω τι γίνεται με τις ελάχιστες διαδικαστικές απαιτήσεις που παρέχουν διαφάνεια, παρέχουν ασφαλεία δικαίου και έτσι μεγαλύπτουμε την παραγωγή, τη θέση σε εμπορία των φαρμάκων, των γενοσύμων και έτσι να ενθαρρύνουμε έρευνα, ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊόντων. Και επίσης ο τελικός στόχος είναι πώς θα έχουμε προσβασιμότητα σε όλους στην Ευρώπη και γι' αυτό τελικά σας διευκρινίζω ότι είμαστε με την πλευρά των εθνικών αρχών, με την πλευρά των ε, καταναλωτών και όχι με την πλευρά της βιομηχανίας. Πρώτα πρώτα θέλουμε πώς θα έχουμε αναβάθμιση της ε, διαφάνειας για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Τώρα όσον αφορά την ε, διαφάνεια θέλουμε να υπάρχει παντού στην λήψη 3, 9, 10, 17, 18, 21, 32, 33 και 38 είναι οι τροπολίες που κατατείνουν προς εκείνο. Η διαφάνεια είναι ε, ένα πάγιο αίτημα πλέον της κοινωνίας όσον αφορά τις τιμές, όσον αφορά την επιστροφή των ε, ιδιωτικών εξόδων για τα φάρμακα και γι' αυτό χρειάζονται και πλέον ε, κάποια μέτρα και θα πρέπει οι αρχές να αποκαλύπτουν, είπαμε, τα τα, τα, τις και για τους ε, ε, εμπειρογνώμονες όπως προαναφέραμε. Αυτό τα λέει η τροπολογία 32. Ε, Άρα θα πρέπει να, είναι, να δημοσιεύονται οι δηλώσεις για συγκρούσει συμφερόντων. Τροπολογία 32. Επίση έχουμε τα, κριτήρια εδώ για, τη, για τιμολόγηση και για ε, τιμολόγηση των σπάντων και επιστροφή εξόδων και, και, το που για 38 επίσης και το πρόβλημα θέμα βάση συμφωνιών συμβατικών για αυτά δεν θα περιλαμβάνονται στη ρύθμιση όμως δεν θέλουμε ευελιξία όμως αυτές οι εξαιρήσεις θα αφορούν κάποιο είδου εκούσιες, συμβάσεων δεν υπάρχει παρακολούθηση, δεν υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία απαιτούν ε, ε, το, το πώς τελικά θα έχουμε κάποια ρύθμιση η οποία θα εξυπηρετεί τους ασθενείς. Τώρα, ε, το ε, τροπολογίες 4 και 14. Ε, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος, όσον αφορά την τιμολόγηση και επιστροφή δαπανών και εδώ είπαμε να υπάρχουν άνετα, άνετα, άνετες προθεσμίες και αυτό σχετίζεται με το τι γίνεται στις περιπτώσεις διασυνοριακών ρυθμίσεων που θα αρχίσουν σε ένα χρόνο. Χρειάζεται όμένω, ένας κοινό ορισμός με κάθε επιφύλαξη των ε, αξιολογήσεων που θα λάβουν χώρα αργότερα. Αυτό θα μας δώσει ασφαλεία δικαίου και θέλουμε έτσι να έχουν ε, συνεπή δράση οι εθνικές αρχές στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Οι εθνικές αρχές δεν πρέπει να φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το HTA γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ομάδες εργασίας και μπορούν οι εθνικές αρχές να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και σε τεχνικό επίπεδο και σε διοικητικό αλλά και όσον αφορά τις συνέπειες των ρυθμίσεων. Τώρα σε σχέση με τις τροπολογίες 6, 7, 8, 35, 36 και 37 οι βασικές διατάξεις εδώ έχουν προταθεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να έχουμε ενημέρωση της ενημερωμένη νομοθεσία κατόπιν της έρευνας του 2009 να μην έχουμε χρειαστές καθυστερήσεις στην αγορά και τέτοιες καθυστερήσεις επίσης να εξεταστεί κατά πόσον ε, θα τηρείται το όριο των 700 ημερών. Κατόπιν τις έρευνες του 2009 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την μη αξιολόγηση των στοιχείων σας παραδείγουμε στο άρθρο 13 και δεν θα πρέπει εδώ σύμφωνα με το άρθρο 14 να έχουμε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Έχουμε αυτή την ρήτρα μία αξιολόγηση. Και ρυθμίζεται ποια, ποιος είναι ο ρόλος των αρχών για τα δεδομένα θέσεως εμπορία και κάποιες άλλες ρυθμίσεις που αφορούν άλλα νομοθετήματα. 15, 16, 20 και 21 τροπολογίες. Εδώ έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τα γενώσιμα σε σχέση με τα ασφαλιστικά συστήματα θα πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη το αν μπορούν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα εθνικές αρχές για τιμολόγηση και επιστροφή εξόδων. Γι' αυτό και σας προτείνω να πάμε στις 25 συν 25 και όχι 15 συν 15 μέρες προθεσμίας. Τώρα, όσον αφορά την ευελιξία των εθνικών αρχών και την ε, αναλογικότητα των προβλεπωμένων μέτρων 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 40 είναι σχετικές τροπολογίες προτείνεται εδώ πέρα η μεγαλύτερη παρέκταση των προθεσμίες για τα φάρμακα νομίζω θα πρέπει να τροπολογήσουμε, να τροποποιήσουν την πρόταση της Επιτροπής για να έχουμε μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των όσων προβλέπονται εδώ. Να μπορούν οι αρμόδιες εθνικές αρχές να έχουν την αυτονομία και την ευελιξία για να συμμορφωθούν με τα όσα επιτάσσει αυτή η οδηγία. Σε σχέση με αυτές τις διατάξεις νομίζω ότι εδώ τα ένδικα μέσα που προβλέπονται με αυτές τις προθεσμίες θα πρέπει να είναι διοικητικού δικαίου όπως προβλέπει το άρθρο 8 και όταν έχουμε δικαιολόγητη καθυστέρηση να, να... ειδοποιούνται διοικητικές και δικαστικές που προβλέπει το Εθνικό Δίκαιο και γι' αυτό εδώ τα σχετικά με οικονομικές κυρώσεις και αποζημιώσεις να απαλληφθούν από εδώ και να γίνουν ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. Το άρθρο 16 επίση λέει για κάποια εθνικά μέτρα τα οποία δεν συμμορφώνονται με την ε, αρχή τη αναλογικότητα και υπερακοντίζουν το σκοπό που έχει θέσει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίση θα πρέπει να έχουμε κάποιε διατάξεις διατάξει όπου θα πρέπει να έχουμε αρκετέ πληροφορίε για να έχουμε την ορθή εφαρμογή της οδηγίας. Γι' αυτό και προτείνω το άρθρο 16 να απαλληφθεί και να δείξουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις εθνικές αρχές. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις. Ήταν πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ που μου ξεκαθάρισαν τις βασικές μας θέσεις. Επίσης, να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία και ιδίω τους ευχαριστώ γιατί έδωσαν το σωστό μήνυμα στο Συμβούλιο και διασκέδασαν τις αμφιβολίες και τους εκφοβιστικούς μύθους που κυκλοφορούσαν και Πάλι ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους καθοδησυγητές και περιμένω προς τη γνώμη τους. Ευχαριστώ πολύ. Και για τις ευχαριστίες προς τη γραμματεία, την οποία καμιά φορά ξεχνάμε όταν ετοιμάζουμε τις εκθέσεις μας, να την ευχαριστήσουμε. Εκ μέρους τώρα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Κούκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαφάνεια είναι κρίσιμη σημασία. Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν βασιζόμενοι στη διαφάνεια και θα εμπιστεύονται τα θεσμικά μας όργανα βάσει της διαφάνειας που μπορούμε να παρέχουμε. Καλώ ορίζω την έκθεση της Κομισιόν και ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά. Μπορώ να υποστηρίξω το... τις περισσότερες προτάσεις του σχεδίου αλλά έχω κάποια άλλα σχόλια, κάποιες προτάσεις και κάποιες αλλαγές να συστήσω. Θα σα εξηγήσω γενικά κάποια από αυτά. Όσον αφορά το εκτιμώντας 15 της πρότασης της Κομισιόν, θα ήθελα να τονίστη το πόσο σπουδαίο είναι τα κράτη-μέλη να μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία κάποιων ε, φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς ε, ή για την εξέταση των διανοητικών δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την πρόταση τη εισηγήτρια να αλλάξουμε το bio-equivalent σε biosimilar, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στι συνέπειες που θα είχε μια τέτοια ενέργεια για τους ασθενείς. Όλοι θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Επίσης, ε, συμφωνώ με την πρόταση της εισηγήτριας ε, ώστε οι διαδικασίες ενημέρωσης και η λήψη αποφάσεων να γίνουν πιο διαφανείς και διαθέσιμες στο κοινό. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τονίσω τις ανησυχίες μου όσον αφορά το εκτιμώντας 15β και το άρθρο 9.2α. Πιστεύω ότι τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων δεν πρέπει να δημοσιεύονται και να καλύπτονται από την αποκάλυψη στοιχείων. Πόση πίεση μπορεί να λαμβάνουν αυτοί οι εμπειρογνώμονες. Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτό αυτό με αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον δεν μπορούμε να δημοσιοποιούμε όλες τις πληροφορίες διότι πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Καλωσορίζω τη φιλοδοξία της εισηγήτριας για παράταση της προθεσμίας για τα γεννόσημα και διαγραφή ορισμένων λεπτομεριών. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να απλοποιήσουμε και να ενοποιήσουμε τα χρονοδιαγράμματα με τα άλλα φάρμακα. Αυτό θα το προτείνω σε πολλές τροπολογίες. Μεγαλύτερη προσβασιμότητα και ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως μεγέθους κράτους μέλους είναι κρίσιμη σημασία. Επίσης, εκτιμώντας, θα ήθελα να αναφέρουμε την, ε, τον ευάλωτο χαρακτήρα ορισμένων μικρών αγορών και την ανάγκη να διατίθενται υποχρεωτικά όλα τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στις λίστες των διεθνών οργανισμών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το εξαιρετικό σας έργο, τη πολύ καλή σας δουλειά, τις εξηγήσεις από την πλευρά της Κομισιόν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, η οποία συνεργάστηκε εξαιρετικά σε ομαδικό επίπεδο για αυτή την οδηγία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση και στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η σκιώδη συγγήτρια από την ε, ομάδα S&D, κυρία Σιλ Τσίλερς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώ την συγγήτρια, την Επιτροπή και τη Γραμματεία μας για την ε, προσπάθεια στην οποία αποδίδονται με αυτό το αυτή την πρόταση νομοθετήματος. Εδώ έχουμε μια πολύ λεπτή ισορροπία να αναζητήσουμε το δικαίωμα δηλαδή των κρατών μελών για την ρύθμιση των θεμάτων δημόσιας υγείας και των σχέσεων με τη φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και την προστασία των ασθενών και την ευρωπαϊκή διάσταση. Βεβαίως θα πρέπει κάθε ασθενής να έχει πρόσβαση σε ε, εν ευθέτω χρόνο κατάλληλη και φθηνή ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν πρέπει κανείς να αποκλείεται λόγω κόστους από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και γι' αυτό καλωσορίζουμε τις αλλαγές της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων προς την τιμή, τιμολόγηση των φαρμάκων με μια καλύτερη προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένε φορέ καθυστερούν στα κράτη-μέλη και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα οι αποφάσει αυτέ ε, όταν πρόκειται μόνο για κράτη-μέλη χωριστά, με επιπτώσει σημαντικέ στον ασθενή και σημαντικέ αποκλήσει ω προ την πρόσβαση στην ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, πράγμα το οποίο θα αντιμετωπιστεί με τη νέα πρόταση. Ωστόσο, θα πρέπει να υπερασπιστούμε και το δικαίωμα των ε, εθνικών αρχών να οργανώνουν όπως το εννοούν το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εσωτερικό τους και βέβαια δεδομένων και των ε, δεινών οικονομικών συνθήκων που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Η οδηγία δεν καθιστά διαφανή την πραγματική τιμή που καταβάλλεται ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόσβαση στα ε, φάρμακα από τον ασθενή. Η μυστικότητα από πλευράς και των αρχών ως προς τις τιμές αγοράς των φαρμάκων και ως προς την πρόσβαση ε, δεν επιτρέπουν ικανοποιητικές συγκρίσεις. Φερρυπίν, στην πατρίδα μου την Ιρλανδία έχουμε καταβάλει τις πιο υψηλές τιμές ανά την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες για φάρμακα και από ό,τι λένε οι εφημερίδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα, ορισμένα φάρμακα υπό δίπλωμα ευρεσιτεχνία ακόμη, τα έχουμε πληρώσει και 50% ακριβότερα από ό,τι το γειτονικό μα Ηνωμένο Βασίλειο. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο βεβαίω. Χωρίς να γνωρίζουμε λοιπόν τι πληρώνουμε, δεν μπορούμε εμείς ή τα κράτη-μέλη να διαπραγματευτούμε ουσιαστικές τιμές. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια και διαπραγματεύσεις για να μπορούν να ελεγχθούν οι τιμές των φαρμάκων. Η ανταλλαγή πληροφοριών μας προς τα τιμολόγια των φαρμάκων έχει κρίσιμη σημασία για να έχουμε καλή και φθηνή πρόσβαση στα φάρμακα. Πρέπει λοιπόν να υποστηριχθεί η βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την οποία αξιοποιούν αρκετά κράτη-μέλη για συγκρίσει τιμών, άλλα μέτρα επίση για την ενίσχυση τη ε, διαφάνεια από τα κρατη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση σε στόχο έχει την ε, γενίκευση των γενοσύμων φαρμάκων με στόχο βέβαια τη συμπίεση προ τα κάτω των προπολογισμών για την αντροφαρμακευτική περίθαλψη κάτω θετικό. Και επίση θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα εγκαίρω να γίνεται και αξιολόγηση τεχνολογικών εξελίσσεων. Ωστόσο, τα, το, τα χρονικά όρια μπορεί να μην υφίστανται ε, σε όρου λογικού για, τα, για όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να δοθούν διαφορετικέ λύσει στη συνέχεια η εισηγήτρια ε, καλώς εισάγει ποινικέ ρήτρε για τα κράτη-μέλη τα οποία δεν τηρούν τις προδιαγραφές και επίσης υποστηρίζω την ε, περάτωση της διασύνδεσης με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, προσπάθεια για περισσότερη διαφάνεια στα κράτη-μέλη και βέβαια προσμένω καλή συνεργασία σε επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ρίβαζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τη συνάδελφα κυρία Παρβάνοβα για την τεράστια δουλειά, το Ηράκλειο έργο που έχει αναλάβει έναντι της οδηγίας αυτής. Έχουμε λοιπόν ε, την ανάγκη για διαφάνεια για τον προσδορισμό της τιμής της, ε, του φαρμάκου. Η πρόταση αυτή της οδηγίας έχει να κάνει με την ε, ταχεία πρόσβαση του ασθενούς στο φάρμακο. Άμα κοιτάξουμε στα πράγματα από πιο κοντά, πρόκειται για λογική φαρμακευτική ανταγωνιστικότητα, η οποία βλέπουμε να έχει επικρατήσει στην όλη αυτή τη διαδικασία. Και γιατί το λέω αυτό, διότι όπως είπε και η το άρθρο 13, το οποίο παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, διότι συμπιέζοντας ε, του προθεσμίες για τον προσδορισμό αναζήτηση και διαπραγμάτευση τιμής για τα νέα φάρμακα, οδηγεί σε ανασφάλεια, οδηγεί σε προβλήματα ως προς την ε, συνθήκες που θα επικρατούν. Γιατί μας λέτε τα κράτη-μέλη θα μπορούν πλέον να επανεξετάσουν, να επαναξελογήσουν την κατάσταση. Κυρία Παρβάνοβα το επισήμανε, το επαναλαμβάνω όμως ότι είναι απαράδεκτο αυτό το επιχείρημα. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητές της όταν προβλέπει δυσανάλογα υψηλέ κυρώσει σε περίπτωση υπέρβαση των προθεσμιών από τι αρμόδιε αρχέ. Είναι υψηλή, ε, είναι πολύ μεγάλη, πολύ αυστηρή η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Είναι πολύ αυστηρέ οι προποθέσει που εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, σε σχέση με την υποχρέωση ενός κράτους, των αρχών ενός κράτους να διαπραγματευτούν νέες τιμές μέσα σε πολύ στο χρονικό διάστημα, ενώ από την άλλη φαρμακοβιομηχανία μπορεί ανά πάσα στιγμή να ψήσει τις τιμές της χωρίς όρια. Αυτό είναι τελείως δυσανάλογο. Άρα λοιπόν, για την ε, τιμή και την αποζημίωση θα πρέπει αυτή να ορίζεται με βάση την προσθεμένη αξία του φαρμάκου. Ξέρετε ότι χώρες όπως η Γαλλία ήδη αναλογίζονται λύσεις διαφορετικές. Σε παραδείγματι να τίθεται μεγαλύτερη αποζημίωση στα φάρμακα εφόσον υπάρχει θεραπευτική προσθεμένη αξία σε σχέση με το νέο φάρμακο που βγαίνει στην αγορά. Και κυρία Περβάνοβα, θα συμφωνήσω ως προς το θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω μάλλον συγκεκριμένα ως προς το θέμα της διευκρίνησης. Θεωρείτε ότι μπορεί να επιτύχει αυτή η λύση, γιατί φαίνεται το Συμβούλιο να αντίκειται στις προτάσεις αυτές. Θεωρείτε ότι μπορούμε να επιτύχουμε και θεωρείτε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα, και εγώ πολύ ευχαριστώ να το κάνω στο πλευρό σας, αλλά θεωρείτε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα για να αναδιαμορφώσουμε 100% την οδηγία αυτή, γιατί αυτή τη στιγμή είναι παράδεκτη. Σε ρωτάω λοιπόν τι πιθανότητες επιτυχίας της οδηγίας αυτής βλέπεις. Πιστεύεις ότι μπορεί να καταλήξει με λύσεις διαφάνειας, δεδομένου ότι υπάρχουν άρθρα το 13, το 16, το 8 που ανέφερες εσύ, που είναι απαράδεκτα στην ε, διαμόρφωση που έχουν αυτή τη στιγμή για τα κράτη-μέλη. Ε, αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί θεωρώ ότι το να αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια για να περάσουμε κάτι το οποίο θα αποτύχει εν τέλει στο Συμβούλιο, ίσως να μην αξίζει τελικά το κόπο. Πρόεδρος. Κύριος Φιέλνερ. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι όσα παρουσιάστηκαν εδώ με βρίσκουν σύμφωνο. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα της διαφάνειας ε, στη διαδικασία τιμής και επιστροφής των φαρμάκων. Ταυτόχρονα αν δεν προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τα επίπεδα τιμολόγησης και επιστροφής. Ε, δεν μου αρέσει όταν έρχονται συνάδελφοι εδώ και κάνω αυτό που πρόκειται να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ αυτό που θα πω τώρα είναι ότι έχουμε ένα σύστημα και σε αυτό το πλαίσιο στη Σουηδία έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα σας δώσω ως παράδειγμα ότι ακόμη και οι καλές προθέσεις μπορεί να κάνουν τα πράγματα άνω κάτω παρότι δεν υπήρχε σκοπός η μόνη μου ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι το πώς ε, σε αυτό το πλαίσιο οι απαιτήσει ε, χρονικών προθεσμιών μπορεί να επηρεάσουν το υπάρχον σύστημα τιμολόγησης και επιστροφής. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, στη Σουηδία, έχουμε ένα σύστημα για τα γενώσιμα που βασίζεται σε έναν μηνιαίο διαγωνισμό τιμών μεταξύ εταιριών και η εταιρεία που κερδίζει και που παρέχει τη χαμηλότερη τιμή ονομάζεται το γενώσιμο του μήνα. Και αυτή η εταιρεία πρέπει να προμηθεύσει όλα τα φαρμακεία όλης της χώρας με αυτό το συγκεκριμένο γενώσιμο φαρμακό. Αυτό κερδίζει κανείς όταν νικάει έναν τέτοιο διαγωνισμό τιμών. Δεν έχω ακούσει κανέναν να επικρίνει τη διαδικασία αυτή. Οι ερευνητές δεν το επικρίνουν. Οι εταιρείε νόσημα φαρμάκων είναι μια χαρά, ικανοποιημένε. Η Επιτροπή δεν έχει παραπονηθεί πότε, διότι πραγματικά υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Και σε μια μικρή χώρα όπως τη Σουηδία εξοικονομεί 700 εκατομμύρια ετησίω αυτό το σύστημα γενώσιμων φαρμάκων. Αλλά αν λέμε ότι έχουμε 15 συν 15 ημέρες ε, στην Κομισιόν, δηλαδή μηνύα ο διαγωνισμό είναι δυνατόν και προτείνεται να αυξήσουμε το προθεσμία 25 συν 25 αυτό το διάστημα, αλλά ούτε αυτό θα το καθιστούσε δυνατό. Δεν θα ήταν δυνατόν να παρέχουν όλα τα φάρμακα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα Παρότι λοιπόν μπορεί να χρειαζόμαστε χρονοδιαγράμματα, προθεσμίες ώστε να διασφαλίζουμε μια διαφανή διαδικασία στα κράτη-μέλη, δεν μπορούμε να την κάνουμε τόσο αυστηρή ώστε να... που να παρεμποδίζει τελικά τα κράτη-μέλη από το να ρυθμίζουν νόμιμα και να οργανώνουν νόμιμα κάτι το οποίο είναι υποτίθεται διαφανές. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που θα συζητήσουμε και περισσότερο με σας κυρία Παρβάνοβα ίσως να υπάρχουν και περισσότερα τέτοια παραδείγματα όπου φιλο... είχαμε τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε διαφάνεια και αυτό παρεμπόδισε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να παρεμποδιστούν και τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ζητώ συγγνώμη που σας μιλάω για ένα εθνικό θέμα, απλά σας έδωσα ένα παράδειγμα άλλων προκλήσεων που γνωρίζω ότι ε, ενέχει αυτός ο κανονισμός. Έτσι γίνεται καμιά φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σκιώδη συγκήτρια τώρα. Κύριε Άλτα Σούσα. Χωρίς μικρόφωνο. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το, και να, ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια η οποία συμπεριέλαβε και τα ορφανά φάρμακα στην έκθεση δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρόταση οδηγίας αυτό το μέτρο είναι εξαιρετικά σημαντικό ώστε να καλύψει κάποια κενά της νομοθεσίας το χρονικό διάστημα δεν είναι δεν έχω πολύ χρόνο συνεπώς θέλω να κάνω τρεις σύντομες ερωτήσεις η έκθεση περιορίζει το πλαίσιο του συμβατικής συμφωνίας, του contractual agreement, κατά κάποιο τρόπο το αποκλείει από την οδηγία και όπως φαίνεται η οδηγία από αυτή την άποψη ουσιαστικά αδειάζει πολιτικά σε σχέση με τις αποφάσεις συμμετοχής στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις στη δική μου χώρα, στην Πορτογαλία. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξή. Πολλά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία έχουν αυτή την τύχη. Ίσως θα έπρεπε να προσθέσουμε κάτι για να επιτύχουμε κάποια συμφωνία. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τα γενώσιμα φάρμακα και την ε, παράταση του διαστήματος από 15 σε 25 μέρες και από 30 σε 50 για την επιστροφή η αιτιολόγηση που δίνεται από την εισηγήτρια έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλα αυτά είναι υποφελή για τις εθνικές υπηρεσίες και για τους καταναλωτές. Θα ήθελα να το εξετάσουμε λίγο καλύτερα. Θα ήθελα κάποιο να μου εξηγήσει τις αιτίε. Υπάρχουν πλέον εκτήματα αν κάνουμε μια τέτοια αλλαγή. Διάφορες εθνικές αρχές ε, θεωρούν το αντίθετο. Θέλω να μάθω συγκεκριμένα σε ποια εθνική αρχή αναφέρεται η συγκήτρια και μετά επαναλαμβάνοντας και τις προηγούμενες ερωτήσεις που ακούσαμε θέλω να ρωτήσω πέρα από το reference product αυτό το προϊόν αναφοράς υπάρχει και μια τιμή αναφοράς για ποιο λόγο δεν μπορούμε να έχουμε μια αυτόματη διαδικασία και για τα γενώσιμα όπως γίνεται ας πούμε για συγκεκριμένες διεθνείς δοκιμές ε, για το Pharmaceutical Inquiry. Αυτό θα επιτρέψει να αποφύγουμε την επανάληψη μιας διαδικασίας που θα μας οδηγήσει σε απολύα χρόνο. Αυτές είναι οι πρώτες μου εισαγωγικές ερωτήσεις σε αυτή την πρώτη συζήτηση. Κάποιες διευκρινήσεις που θεωρεί σημαντικές η ομάδα μου. Να μας δώσει. Η Ευχαριστώ. Köszönöm Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είναι εξαιρετική η έκθεσή της. Συμφωνούμε στα περισσότερα με όσα είπε. Είναι πολύ σημαντικά όσα μας εξήγησε στην εισηγήσή της. θέλουμε να ενεργούμε για το συμφέρον των ασθενών και όχι της βιομηχανίας. Και εμείς εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους, αλλά και τους Ούγγρους βέβαια, Έχουμε αυτές τις προτάσεις ε, υπάρχουν κάποιε προτάσει τροπολογιών επί του κειμένου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε δεν βοηθούν όσον αφορά τα ε, γενώσιμα, όσον αφορά λοιπόν το πώ θα είναι πιο αποτελεσματική θέση εμπορία του. Και συμφωνώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε να αποτελέσουμε, να επιτελέσουμε δηλαδή το πώ θα έχουμε αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Αυτέ οι 15 μέρε που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα χρονικό διάστημα πολύ σύντομο. Ελπίζω ότι η πρόταση της κυρίας Παρβάνου για 25 μέρες, συν 25, ε, θα θεωρηθεί πιο ευέλικτο στην πράξη. Και εμείς θα αποδειχθούμε πιο ευέλικτοι στην πράξη. Τώρα, κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε κάποια πρόταση, η οποία θεωρούμε ότι είναι ένα πίσω γύρισμα όσον αφορά την τιμολόγηση την πιο διάφανη που θέλουμε. Γιατί, γιατί τα κράτη-μέλη πάντοτε θα πρέπει να παρέχουν για την τιμολόγηση πληροφορίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχουμε το σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο είχαν συμμετάσχει 18 κράτη-μέλη. Και η Ουγγαρία είχε συμμετάσχει και βρισκόμαστε άνω του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε συγχρηματοδοτήσει κατά 19%. Πληρώσαμε 8,5% οι αυστριακές ε, αρχές, ένα 0,5% όσον τα λειτουργικά έξω του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό και ήταν πάρα πολύ καλό, μια που όλα τα κρατημέλη μπορούσαν να πληροφορηθούν την τιμολόγηση των φαρμάκων σε άλλες χώρες. Άρα υπήρχε συγκρισιμότητα, μπορούσε κανείς να έχει επιχείρημα προς τις φαρμακοβιομηχανίες, βοήθησε πάρα πολύ και τελικά ωφελήθηκαν οι καταναλωτές γιατί δεν μπορούσαν να βρούνε τα φάρμακά τους σε καλές τιμές. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η πρόταση αυτή είναι αξιόλογη. Την υποστηρίζουμε. Τώρα το άρθρο 16 κυρία Παερβάνοβα και η προτινόμενη διαγραφή του. Νομίζω δεν χρειάζεται αυτό το άρθρο. Δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε κάτι και γι' αυτό το πιο σωστό είναι το άρθρο αυτό να απαλληφθεί. Το άρθρο 18 θα μας λύσει το πρόβλημα για ένα τμήμα τέλο πάντων. Το άρθρο 16, εάν δεν το απαλείψουμε, αυτό θα αποτελέσει υπερβολή κάτι το περίτω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κύριε Λεπάζου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ και να συγχαρώ την κυρία Παρβάνοβα και για την πολύ ογκώδη δουλειά που έχει αναλάβει. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ε, συμπερίληψη των νομοθετικών της παραπομπών στις αιτιολογικές σκέψεις που έτσι καθιστούν το έργο πολύ πιο σαφές. Πολύ σημαντικό είναι το, η κατάργηση του συστήματος κυρώσεων για μη τήρηση των προθεσμιών. Πολύ καλά κάνει δηλαδή και ξεκαθαρίζει από τα θέματα αυτά το άρθρο 8 εισηγήτρια. Αλλά επίση δεν θέλω να αναφερθώ σαν συμπληρωματικό επιχείρημα σε αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Πού βρίσκονται αυτέ, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την δυνατότητα χρηματοδότηση των συστημάτων υγεία. Επίση, η εισαγωγή ενό νέου άρθρου για τη διαφάνεια και τη συγκλού συμφερόντων είναι πολύ σημαντική. Ε, για τα γενώσιμα, η ενίσχυση των προθεσμιών έχει σημασία για τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και για τον ασθενή. Ωστόσο, οι 15 συν 15 μέρες Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ε, προϋπόθεση για χωριστή αξιολόγηση κάθε προϊόντος είναι πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και καλά κάνει η συζήτρια για να, που προτείνει επιπλέον περιθώριο χρονικό. Για να συμφωνήσω με την κυρία Ριβαζή θα ήθελα να πω ότι είναι μάλλον ε, επίοικης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκθεση ως προς τα υπόλοιπα των φαρμάκων. Ε, δεν είναι αποδεκτές οι προτάσεις στις 20 ημέρες. Άλλωστε δεν είναι αποδεκτές και για τα κράτη-μέλη η διαδικότητα της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας επιπλέον ενισχύει το περίπλοκο χαρακτήρα των μέτρων. Θα πρέπει λέει, τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ποιότητα μαζί με την προϋπόθεση της αποζημίωσης και έτσι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστω και με τροποποίηση της εισηγήτριας, μου φαίνεται όχι καλά διατυπωμένη, δεν είναι καλά ισορροπημένη και ω εκ του δεν ότι θα εγκριθεί από το Συμβουλίο. Και γι' αυτό έρωτα την κυρία Παρβάνοβα και εγώ ποια θεωρεί ότι είναι η καταλληλότερη στρατηγική, ποια θεωρεί ότι είναι η στρατηγική που πρέπει η Επιτροπή μα να υιοθετήσει, η συγγήτριά μα να προωθήσει προκειμένου να εξασφαλίσουμε την έγκριση του κειμένου εν τέλει και από το Συμβούλιο για να πάει προς την κατεύθυνση που εμείς επιδιώκουμε, όπως άλλωστε και η ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την κυρία Λεπάζ και τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει πολύ την εισηγήτρια για τα όσα με σαφήνεια μας εξήγησε από την πρότασή της. Σύμφωνα με τους στόχους και με το πνεύμα του κειμένου πρόκειται για μια οδηγία 22 ετών που χρήζει ανακαίνηση. Έχει αλλάξει η αγορά στο μεταξύ, οι εθνικές πρακτικές και έχει αλλάξει και το σχετικό δίκαιο. Άρα, θέλουμε εξυγχρονισμό τώρα της ρύθμισης. Πρώτα πρώτα, για να είναι πιο ανταγωνιστική η βιομηχανία όσον αφορά τα διοικητικά. Δεύτερος λόγος είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς εύκολα και γρήγορα θα έχουν πρόσβαση στα φάρμακα. Τρίτο λόγο. είναι να έχουμε εξοικονόμηση δαπανών μια που περνάμε κρίση οικονομική. Άρα μπορούμε έτσι να πετύχουμε τους στόχους μας. Από της πλευράς. Επίσης, αυτή η οδηγία λαμβάνει υπόψη την αρχή της επικορικότητας. Μια από πρότασή μας αφορά μόνο διαδικαστικούς κανόνες. Δεν θέλουμε να ενεργονίσουμε ούτε επιστροφή εξόδων, ούτε την τιμολόγηση. Προσπαθούμε απλώ να προσαρμόσουμε την νομοθεσία μας στην πραγματικότητα. Τώρα, να σταθώ στα όσα άκουσα. Πολύ ενδιαφέρον στις να μην υπάρχει επικάλυψη των διαδικασιών. Δεν θέλουμε να μην μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση τα κρατημέλη όταν όσο έχουν ήδη αξιολογήσει αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μην έχουμε τις ίδιες αξιολόγησεις επικάλυψη. ούτε θέλουμε να έχουμε εδώ εμπλοκή των δικαιωμάτων της πνευματικής διοκτησίας. Για τα γενώσιμα, για τα φάρμακα που κανονικά εύκολα μπορεί να τα βρει κανείς. Κάτι άλλο επίσης όσον αφορά τα γενώσιμα θέλουμε να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση και σε πολλές χώρες με την ρύθμισή μας θα έχουμε μεγάλες οικονομίες για τον προπολογισμό. Να επομένως, γιατί όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τον εθνικό προπολογισμό. Ευχαριστούμε επομένως όλους όσους έχουν τον λόγο και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ληφθούν υπόψη όλα όσα έχουν προταθεί και από το Συμβούλιο να καλύψουμε επομένω έτσι τις ανησυχίες των κρατών μελών. Θα λάβουμε όλο όσα είπατε υπόψη. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια για την πρωτεία του Συμβουλίου γιατί εντατικά εξεργάζεται αυτή την πρότασή μας. Ευχαριστώ πολύ και για να κλείσουμε τώρα σε ακούσουμε την εισηγήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους και τους συγκεκριτές, όλους τους συναδέλφους που μοιράστηκαν μαζί μας τις απόψεις τους για αυτό το θέμα, το περίπλοκο. Πολλά θέματα χρήζουν διευκρίνησης με τα κράτη-μέλη και θα ήθελα να αναφερθώ στις πολιτικές Συνεπής ε, και την ε, πιθανότητα της πολιτικής επιβίωσης αυτού του νομοθετήματος, τα ζητήματα δηλαδή που έθιξε η κυρία Ριβαζή πρώτη. Καταρχάς, ξεκινάμε από σημείο απόλυτου παγώματος, λόγω της, των δισταγμών των κρατών. Εγώ προσπαθώ να ανοίξω το πεδίο. Ε, άλλαξα πολλά πράγματα, άλλαξα πολλά πράγματα στην πρόταση της Επιτροπής ιδιαίτερως, διότι θεωρώ ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι κρίσιμο να μην εκτεθούν τα κράτη-μέλη σε περαιτέρω πιέσεις και ιδιαίτερα οικονομική αβεβαιότητα. Αλλά όχι και να αλλά ούτε και να γίνει πιο δύσκολη η δουλειά ε, και οι διαδικασίες για τις εθνικές αρχές να τις οδηγήσουμε σε πτώχευση. Χρειάζεται περισσότερη βεβαιότητα, περισσότερη προβλεψιμότητα και διαφάνεια και καλύτερη πρόσβαση για τον ασθενή σε καλύτερα φάρμακα, σε πιο οικονομικά φάρμακα. Γι' αυτό λοιπόν, αφού κοιτάμε τα αποτελέσματα από την έρευνα στον τομέα του 2009 και τα συμπεράσματα που καταγράφονται σε αυτή την μελέτη, για τον τομέα, είναι απόλυτος απαραίτητο να κλείσουν ε, οι... να αλλάξουν οι ρυθμίσεις, όχι μόνο λόγω των εξελίξεων, αλλά και γιατί είναι πολύ δύσκολη η εποχή που διέρχονται οι κυβερνήσει και τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες πολύ αδιαφανείς και συμφωνώ με τον κύριο Φιέλνερ ότι η κατάσταση του κάθε κράτους μέλους πρέπει χωριστά να αξιολογείται και εγώ βεβαίως πολύ ευχαριστώ θα συζητήσω με τους συναδέλφους, με τους και ηγητές ε, λεπτομερώς για να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προστέψουμε τις εθνικές αρχές από αδικαιολόγητες πίεσεις ταυτόχρονα όμως προστατεύοντας και τον ασθενή από αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, και την υποχρέωση να το πράξουμε για, την, ε, για τα βιοεισοδύναμα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα γενώσιμα δηλαδή. Η βιοομοιότητα, biosimilarity, έχει να κάνει με παρόμοια προϊόντα που επίσης έχουν, λάβει, έχουν αδειοδοτηθεί. Πνευματική ιδιοκτησία, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η τομεακή έρευνα δείχνει αδιαφυσβήτητα στοιχεία πως Έχουν γίνει κάποιε προσφυγέ για παραβίαση πνευματική ιδιοκτησία κατά τρόπο καταχρηστικό και θα πρέπει αυτό να εμποδίζεται. Επίση, για τη θεσιμότητα των πληροφοριών, γιατί προσπαθώ να, προσπαθώ να δώσω στο το του ευελιξία στα κράτη-μέλη, μεν, αλλά για του εμπειρογνώμονε, για τη διαφάνεια. Ύστερα από όλε αυτέ τι συζητήσει, εάν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλει να ανοίξει τις ε, πόρτες της ε, διαφάνειας, θα πρέπει και να το πει δημόσια στην κοινή γνώμη. Η συζήτηση, όπως τη βλέπω, προτείνει μάλλον προς ε, απαιτήσει για περισσότερη διαφάνεια, για περισσότερη κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων. Προσθέμενη αξία. και δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικά εθνικά συστήματα. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει να εξασφαλιστεί η ισορροπία, δικαιοσύνη, είναι το να ε, χρησιμοποιηθεί το HDA γιατί στηρίζεται σε στοιχεία, πραγματικά. Κάθε τι άλλο θα ήταν αυθαίρετο. Ένα σύστημα όμω ενιαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσέφερε και περισσότερη διαφάνεια και πιο ισόρροπη αντιμετώπιση. για την επιδίωξη και συμπίεση των τιμών και το όφελο από την εισαγωγή των γενοσύμων. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δίνονται αποδείξει ότι, ότι μειώνει την ε, τιμή των φαρμάκων η εισαγωγή γενοσύμων ή ότι βελτιώνει την πρόσβαση για τον ασθενή. Μου φαίνεται δεδομένο. Βεβαίως, κατά άλλα, ε, ε, ακολουθούμε πάντοτε την αρχή της ε, την αρχή ότι τις τιμές τις ορίζουν τα κράτη-μέλη. Επιδιώκουμε βεβαίως εναρμόνιση όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά πάντοτε θα γίνεται παραπομπή στην Εθνική Αρμόδια Αρχή. Εν γέννη. Εγώ θέλω την βέλτιστη δυνατή συνεργασία με τους ε, συναδέλφους, ιδιαίτερα τους Κιώδης, για να προχωρήσει το θέμα αυτό που πιστεύω θα είναι προς όφελος των πάντων και έχουμε μια σειρά κρατών μελών που διστάζουν ακόμη και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσφέρουμε την υποστήριξή μας στην Κυπριακή Προεδρία για τις προσπάθειές της να διευκρινίσει αλλά και να πείσει τα κράτη-μέλη ότι αυτό που πράττουμε μόνο για να τους, τα βοηθήσουμε γίνεται, για να τα στηρίξουμε στην επιδίωξη καλών διαφανών ε, λύσεων. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ την Συγκητρία. «19 Οκτωβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες, 12 το μεσημέρι. Μαζί με τις τροπολογίες στις 28 Νοεμβρίου συζητούμε πάλι την έκθεση εδώ για να την εξετάσουμε, να την ψηφίσουμε δηλαδή στις 18 Δεκεμβρίου εδώ στην Επιτροπή και για την Ολομέλεια δεν έχουμε ακόμη προθεσμία. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και πάλι, για τη δουλειά σας, για τη στράτευσή σας. Και προχωρώ στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. 6 διορθώνει ο μιλητής. Προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρήπανση, δυστυχώς. Η συγγετρία δεν μπορεί να είναι εδώ, ούτε και οι σκιώδεις συγγετές. Συγγνώμη ένα λεπτό, λέει ο πρόεδρος. Er- Α, όχι, δύο είναι εδώ, μάλιστα, ο κύριος Σαταρέλα και ο κύριος Κυλακάκης. Τότε ας ακούσουμε τους σκιώδεις συγγετές. Αν δεν μπορεί η κυρία Ρόσπαχ να βρει αντικαταστάτη στην ομάδα της, ας ακούσουμε τους σκιώδεις συγγετές. Τον κύριο Ταταρέλα πρώτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τη συναδελφό Ροσμπαχ για την έκθεση και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει την προσχωρήση στο πρωτόκολλο. Αυτή η επικυρώση έρχεται αργά και είναι το πρώτο βήμα για μια ισχυρή συνεργασία με τις υπόλοιπε χώρες ε, στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Χωρίς κοινή πολιτική μεταξύ όλων των χωρών της Μεσογείου δεν θα είναι δυνατή η προστασία ε, της, Μεσογείου. Η καταστροφή στον κολπό του Μεξικού το 2010 έδειξε ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες δεν παρουσιάζουν καμία ασφάλεια. Ειδικότερα όταν πραγματοποιούνται σε μεγάλα βάθη. μια διαρροή υδρογονανθράκων όπως το 2010 σε μια ημίκλειστη θάλασσα όπως είναι ο Σόγιος θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες και ε, οριστικές συνέπειες ε, μη αναστρέψιμες για τους θαλάσσιους οικοτόπους αλλά και για την οικονομία των χωρών που βασίζονται στον τουρισμό και στην αλληλεία. Θα πρέπει δηλαδή να λάβουμε υπόψη ότι η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί ένα μοναδικό στον κόσμο φυσικό περιβάλλον, η ευημερία του οποίου εξαρτάται από την προστασία των φυσικών του πόρων και από τη σπουδαιότητα των τουριστικών του δραστηριοτήτων. Αυτούς τους μήνες ε, στην Ιταλία λαμβάνει η χώρα μια ισχυρή κινητοποίηση κατά των εγκρίσεων που έχουν ήδη εκχωρηθεί από, την Ιταλική, από το Ιταλικό κράτος ε, για την Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα κοντά στις νήσους Τρέμητη που σημειώνω αποτελούν ένα προστατευόμενο περιβάλλον το οποίο πρέπει να προφυλαχθεί με οποιοδήποτε κόστος. Η επικύρωση του πρωτοκόλου συμπληρώνει την νομοθετική πρόταση Παράλληλα με την επικύρωση του πρωτοκόλου, χθε ψηφίστηκε στην Επιτροπή Ήτρε η οδηγία για την ασφάλεια των υπερακτήων δραστηριοτήτων που ανεβάζει τα πρότυπα ασφαλεία για τις ερευνητικέ διαδικασίες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τις ρυθμίζει και επιτρέπει τον παροπλισμό μια εγκατάσταση δημιουργεί σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος, αυξάνει την ευθύνη των φορέων και ενισχύει τη σπουδαιότητα της αξιολόγησης του κινδύνου και της ε, δημόσιας συμμετοχής ε, στην έγκριση υπερακτών δραστηριοτήτων. Δυστυχώς, οι συνάδελφοί της Επιτροπής Ήτρε προτίμησαν την οδό της οδηγίας αντί για ε, τον πιο γρήγορο κανονισμό είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί αυστήρα η συνθήκη. Γι' αυτό το, λίγα, γι αυτό το λόγο οι άδειε πρέπει να δοθούν μόνο σε φορείς με οικονομικές και τεχνικές ικανότητες τέτοιες που να μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των υπεράκτων δραστηριοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να συντάξουν εκθέσεις που να περιλαμβάνουν εκτίμηση κινδύνων και σχέδιο Έκτακτη ανάγκης πριν ξεκινήσουν τις δραστηριότητε Σε αυτό το πλαίσιο ακόμη και οι εθνικέ αρχές παίζουν ε, σημαντικό ρόλο στην ευθύνη των ελέγχων ασφαλείας. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει γέτιδα στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στην Μεσόγειο με όλο και πιο αποφασιστικές συμφωνίες ε, επικεντρωμένες στην προστασία της Μεσογείου. Ευχαριστώ κύριε Τερέλα. Ας ακούσουμε τώρα τον σκιώδη συγκητή εκ μέρους των φιλελευθέρων, τον κύριο Σκυλακάκη. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. President. This protocol... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το πρωτόκολλο είναι παλιό, αλλά περιλαμβάνει τη συνθήκη της Βαρκελόνης που είναι μια ικανή διαδικασία για τη διεθνή συνεργασία στη Μεσόγειο. Για εμάς ε, στη Μεσόγειο όπου ο τουρισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για τις οικονομίες ε, του Ιταλικού Νότου που διαρχείται περίοδο κρίσης. Η προστασία της Μεσογείου είναι εξαιρετικά σημαντική. Μιλάμε για προστασία όχι μόνο από τι δικέ μα δραστηριότητε. Θα μπορούσε αυτό να αντιμετωπιστεί με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μιλάμε και για τις δραστηριότητες άλλων μεσογειακών χωρών. Αποδεχόμενοι αυτό το πρωτόκολλο, όπου θα συμμετέχουν και άλλε χώρε τη Μεσογείου, παρέχουμε στην Κομισιόν ένα εργαλείο ώστε να προχωρήσει και να πείσει όλες τις χώρες της Μεσογείου να αποδεχθούν και να συμμετέχουν σε αυτό το πρωτόκολλο. Δεν είναι το καλύτερο πρωτόκολλο που θα μπορούσε να υπάρχει, είναι λίγο παλιό, αλλά πιστεύω ότι αν γίνει δεκτό αυτό το πρωτόκολλο θα παρέχει ελάχιστα τουλάχιστον πρότυπα. Αυτό ουσιαστικά είναι μια άσκηση εξωτερικών σχέσεων. Το υποστηρίζω λοιπόν και ελπίζω ότι η Κομισιόν θα ε, χρησιμοποιήσει σωστά την ψήφα μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαπρός έχει το λόγο. Ναι, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Υποστηρίζω απόλυτα τα όσα ε, είπε ο κ. Σκυλακάκης. Είναι παλιό πρωτόκολλο. Αξίζει να υπάρχει και να υπογραφεί από ορισμένους από τους εταίρους μας στη Μεσόγειο. Έχει ήδη επικυρωθεί από την Αλβανία, την Τινησία, το Μαρόκο, τη Λιβύη, την Κύπρο και τη Συρία. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να το επισημάνει αυτό, να το υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να ελπίζουμε. Πρέπει να το προσαρμόσουμε στο κείμενο που συζητάτε αυτή τη στιγμή, για το οποίο αποφασίσαμε πριν από λίγο καιρό σε σχέση με τις ε, υπεράκτιες εγκαταστάσεις, πλατφόρμες, ε, Συμμερίζομαι την ανησυχία για τους κινδύνους ε, των υπεράκτιων ε, εγκαταστάσεων στη Μεσόγειο που υπενθυμίζω η Μεσόγειος ανανεώνεται μόνο κάθε 100 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο όπως η Μάγχη για παράδειγμα ή ο Ατλαντικός. Έτσι λοιπόν ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη διασφάλιση της εκμετάλλευσης των θαλασσών μας ε, είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπογράψουμε αυτό το πρωτόκολλο παρότι δεν πρέπει να είμαστε αγαθοί και να νομίζουμε ότι θα λύσουν όλα μας τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πλευρά της Κομισιόν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο για τη δουλειά που έχει κάνει και για την υποστήριξή του. Θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Είναι απαραίτητο και επίγον να επικυρώσουμε αυτό το πρωτόκολλο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο διότι θα αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο προστασίας της Μεσογείου από ατυχήματα ε, και ρήπανση με πετρέλαιο από υπερακτές δραστηριότητες, αλλά όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, γιατί θα αποτελέσει ένα πολιτικό μήνυμα προς τους εταίρους μας στον Νότο, ώστε να συντονίσουμε τις προσπαθίες μας και να ακολουθήσουμε να συνεχίσουμε αυτή την, ε, ε, το συνολικό εγχείρημα προστασίας της Μεσογείου από τις υπεράκτητες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας για σήμερα το πρωί. μια συζήτηση για τις τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε τα απόγευμα. Κατά πάσα πιθανότητα πάμε για την πρώτη ολομέλεια του Νοεμβρίου με το θέμα αυτό. Σας εύχομαι. Καλό μεσημέρι, καλή όρεξη σε όλους. Πάρτε δυνάμεις για να ξαναρχίσουμε όπως πάντα στις 3 ακριβώς με τις προθορίες είστε δεν είστε.